Αγαπητοί ε, προσκεκλημένοι, αγαπητοί ομιλητές, με μεγάλη τιμή κηρύσω την έναρξη της ε, συνεδρίασης της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής επ' ευκαιρία της Διεθνούς ημέρας της Γυναίκας του 2019 για την ε, εξουσία των γυναικών στην πολιτική. Με μεγάλη χαρά θα σας παρουσιάζω σήμερα 23 μέλη από 16 εθνικά κοινοβούλια και την Νορβηγία – σας καλωσορίζω όλους και θα ακούσουμε ενδιαφέρον την συνεισφορά σας σε αυτή τη σημαντική συζήτηση. Καταρχάς, θα ήθελα να κάνω λίγες πρακτικές ανακοινώσεις. Η εκδήλωση σημερινή οργανώνεται σε συνεργασία με την Διεύθυνση για τις σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Η διερμηνία υπάρχει σε όλες σχεδόν τις ε, γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εξαίρεση των Ιρλανδικών. Η συνεδρίαση μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Κατά τη διάρκεια της έναρξης της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να πάρουν τον λόγο. Θα έχουν την ευκαιρία όμως να μιλήσουν κατά τη διάρκεια των πάνελ. Επίσης, σημειώστε ότι ο χρόνος για τις παρεμβάσεις από τους ομιλητές των πάνελ και από το κοινό είναι περιορισμένος. Θα υπάρχει χρονομέτρηση κατά τη διάρκεια των ομιλιών, ούτως ώστε να παρακολουθεί ο καθένας τον χρόνο. Αν θέλετε να ζητήσετε το λόγο, τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων μπορούν να συμπληρώσουν ένα από τα έντυπα που μοίρασαν οι κλητήρε, οι οποίοι θα τα συλλέξουν αυτά τα έντυπα μετά. Και αν είσαστε χρήστες του Twitter, το hashtag για, το, για τη σημερινή εκδήλωση είναι Women's Power and Politics. Και τώρα θα δώσω το λόγο για την αρκτήρια ομιλία στο προ πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντώνιο Ταγιάννη. Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Λίχα. Πρόεδρε της Κροατίας, της Δημοκρατίας της Κροατίας, Δημήτρη Παπαδημούλη. Και προσκεκλημένοι μας, με μεγάλη χαρά έρχομαι εδώ ενώπιόν σας μία μέρα πριν τη Διεθνή ημέρα της γυναίκας για να εκδηλώσουμε τα πιο σημαντικά πρόσωπα στη ζωή μας, τη μητέρα μας, τις αδερφές μας, τις ξαδέρφες μας, τους φίλους, τις φίλες μας. Σήμερα υπάρχουν, ακόμα και σήμερα, τρομερές διακρίσεις εναντίον των γυναικών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ευρώπη είναι μία από τις πιο ευημερούσες και πιο ελεύθερες περιοχές του κόσμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, εξασφαλίζει τις πιο ισότιμες κοινωνίες για άνδρες και γυναίκες. Οι ίσες ευκαιρίες είναι πυλώνας για την πρόοδο της κοινωνίας μας. Πρέπει να συνεχίσουμε όμως τις προσπάθειες, γιατί έχουμε πολλά ακόμα να επιτύχουμε σε πολλούς τομείς. Η ισότητα, καταρχάς, σε θέματα ελευθερίας, ελευθερία να επιλέξει κανείς το μέλλον του, να σπουδάσει, να δουλέψει και να είναι ελεύθερος από οποιοδήποτε στερεότυπο. Υπάρχουν πολλοί αριθμα δικαιώματα που υπερασπιζόμαστε. Θυμάμαι την απόφασή μου. Κατά την απόφαση εναντίον του συναδέλφου Κόρβι Μίκελ, μετά από την αδιανόητη ομιλία στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο έπαιξε πάντα σημαντικό ρόλο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως στην απελευθέρωση της Άζια Μπίμπη ή στην απονομή του βραβείου Σαχάροφ σε θραλές γυναίκες τη Μαλάλα Σαφουσάη, την Άντια Μουράτ και τη Λάμια Μπασάρ. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τιμήσουμε τη Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίσια, την θαραλέα αυτή δημοσιογράφο που σκοτώθηκε στη Μάλτα πριν από ένα χρόνο ακριβώ. Θέλουμε να μάθουμε το όνομα όχι μόνο των δολοφόνων, αλλά και των οικογενειών των δολοφόνων. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βάλουμε περισσότερες γυναίκες στην πολιτική, σε υψηλές θέσεις, καθώς και στον επιχειρηματικό κόσμο. Δεν είναι μια μάχη μεταξύ ανδρών και γυναικών αυτή. Είναι μια μάχη για μια ισχυρότερη Ευρώπη που δεν μπορούμε να την πετύχουμε χωρίς την πλήρη αναγνώριση των δικαιωμάτων των γυναικών και είναι μια μάχη υπέρ της αξιοπρέπειας και της ασφάλειας όλων. Χρειαζόμαστε γυναίκες στην εξουσία, χρειαζόμαστε γυναίκες στην πολιτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε Αντώνιο Ταγιάννη για την ε, ενακτήρια αυτή ομιλία και τώρα ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Παπαδημούλης, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που ήρθατε στην εκδήλωσή μας. Είναι μια πολύ σημαντική συνεδρίαση αυτή. Μία μέρα πριν από τη Διεθνή Μέρα της Γυναίκας, 80 μέρες πριν από τις ε, ευρωεκλογές και θα μιλήσω ως αντιπρόεδρος υπεύθυνο για την ισότητα και την ποικιλομορφία και θα περάσω στην μητρική μου γλώσσα, τα ελληνικά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σας. Είμαι χαρούμενος γιατί βλέπω τόσο μεγάλη συμμετοχή ε, και ε, από πολλές χώρες και θέλω να σας πω μερικές ιδέες σύντομα για το τι έχουμε κάνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, για να προωθήσουμε την ισότητα αυτά τα τελευταία πέντε χρόνια όχι μόνο ως αρμόδιος αντιπρόεδρος αλλά και ως πολίτης που εστερνίζομαι αυτές τις αξίες, τις ισότητες. Πιστεύω ότι για να μπορέσουν οι γυναίκες να διεκδικήσουν έμπρακτα και να πετύχουν την ισότητα, χρειάζεται να τους δοθεί η δυνατότητα να είναι πιο ορατές, να έχουν πραγματικά ίσες ευκαιρίες, έτσι ώστε να πετύχουν ορατή εκπροσώπηση. Στο Ευρωκοινοβούλιο έχουμε πολλές γυναίκες που είναι πρόεδροι ή συμπρόεδροι πολιτικών ομάδων, που είναι πρόεδροι επιτροπών. Άρα στο σκέλος Women in Politics έχουμε μια επαρκή εκπροσώπηση. Αλλά αν δούμε τις κορυφές, θα δούμε ότι στην κορυφή όλων των ευρωπαϊκών θεσμών έχουμε άντρες. Άνδρας πρόεδρος στο Συμβούλιο, άνδρας πρόεδρος στην Κομισιόν, άνδρας πρόεδρος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άνδρας πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, άνδρας πρόεδρος στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, άνδρας πρόεδρος στην Επιτροπή Περιφερειών. Δεν υπάρχουν γυναίκες που να μπορούσαν να είναι κατάλληλες για κάποιες από αυτές τις προεδρίες. Η γνώμη μου είναι ναι. Και ελπίζω οι επόμενες ευρωεκλογές να βοηθήσουν μαζί με τις συζητήσεις που θα γίνουν μετά τις ευρωεκλογέ, έτσι ώστε σε κάποια από αυτά τα κορυφαία πόστα να έχουμε και γυναίκες. Δεύτερη παρατήρηση. Σήμερα είμαστε σε ένα πάνελ όπου η πλειοψηφία είναι γυναίκες. Αλλά αυτό είναι δυστυχώς η μικρή εξαίρεση, η σπάνια εξαίρεση. Συνήθως τα πάνελ στις δημόσιες συζητήσεις είναι ανδροκρατούμενα. Και πρέπει και αυτό να αλλάξει και χαίρομαι γιατί η Επίτροπος Γιούροβα μετέχει σε μια πρωτοβουλία για να αλλάξει αυτό το πράγμα διότι αν δεν υπάρχει ορατότητα μεγαλύτερη για τις γυναίκες που μετέχουν στα κοινά ε, θα δυσκολευτούν περισσότερο να κατακτήσουν θέσεις που τους αξίζουν. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό την Προεδρία μου έχουμε συγκροτήσει ένα ε, high-level working group, το οποίο ετοίμασε, ενέκρινε ομόφωνα και υιοθέτησε ομόφωνα και το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ένα πλάνο να ενισχύσουμε την ισότητα στην πράξη μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάναμε κάποια βήματα θετικά. Ας πούμε για παράδειγμα, μέσα στο 2018 το 58% των νέων head of units είναι γυναίκες. Στο επίπεδο το μεσαίο της διοίκησης αυξήθηκε από το 30% στο 40% η παρουσία των γυναικών ως επικεφαλής μονάδων διοίκησης. Στο επίπεδο των γενικών διευθυντών κάναμε επίσης μια πρόοδο και έχουμε φτάσει, είχαμε βάλει στόχο να φτάσουμε στο 35%, είμαστε στο 34% πολύ κοντά αλλά στους γενικούς διευθυντές που είναι η κορυφή της διοίκησης το ποσοστό των γυναικών είναι κάτω από 20%. Πράγμα που σημαίνει ότι όσο πλησιάζουμε προς την κορυφή ο στόχος της ισότητας αδυνατίζει. Πετύχαμε να υιοθετηθεί και ένα σχέδιο για μια ουδέτερη ως προς το φύλλο γλώσσα. Έχουμε κάνει βήματα για την αντιμετώπιση του harassment και μέσα στο Κοινοβούλιο σε συνεργασία και με το κίνημα MeToo που υπάρχει και μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε κάνει μια πρόοδο, αλλά μένουν πολλά να γίνουν. Τελειώνω με έναν αριθμό. Σύμφωνα με μια μελέτη του ΟΗΕ, αν συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς, θα πετύχουμε την πλήρη ισότητα των δύο φύλων σε 182 χρόνια. Είναι πολύ αργά για να συνεχίσουμε να κινούμαστε με τέτοιου ρυθμούς πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητα. Και αυτό οφείλουμε να το κάνουμε όχι μόνο οι γυναίκες που είναι στην πρωτοπορία αυτού του στόχου, αλλά και οι άνδρες που συμμερίζονται αυτές τις αξίες, γιατί η ισότητα ανδρών και γυναικών είναι πριν απ' όλα θέμα δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Ευχαριστούμε για την ομιλία σας. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κροατίας, η κυρία Γκραμπάρ Κιτάροβιτς, θα κάνει τη σημερινή της ομιλία. Είναι από τις πιο γνωστές γυναίκες πολιτικούς. Είναι σημαντική αυτή η θέση που έχει, γιατί έτσι βλέπουν και οι νέες γενιές ότι οι γυναίκες μπορούν να τα καταφέρουν όλα. Η κυρία Κολίνα, Κολίντα Γκράμπαρ Κιτάροβιτς, πρόεδρος της Κροατίας, θα μας βγάλει την ομιλία της. Mr. Uh, πρόεδρε του Κοινοβουλίου, ε, κυρία Επίτροπε, πρόεδρε της Επιτροπής ΦΕΜ, ε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων, κυρίε και κύριοι. Αποτελεί μεγάλη μου χαρά το να βρίσκομαι σήμερα εδώ για να παρέμβω στο πλαίσιο της σημερινής εκδήλωσης ε, στα πλαίσια της ε, Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας. Ε, θεωρώ ε, πως η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γενικών και των φιλοδοξιών τους αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες μας πολίτερα του κόσμου και της Ευρώπη ως ε, πρώτη πρόεδρος ε, της ε, Κροατίας βρίσκομαι ενώπιον σας και βέβαια αυτό αποτελεί μια ένδειξη ως προς το πώς έχουν τα πράγματα, αλλά δεν αποτέλεσε κάτι το αυτονόητο. Χρειάστηκε να επιμείνω έτσι ώστε να διεκδικήσω αυτή τη θέση. Και χρειάστηκε να κάνω πολλές υπερβάσεις ε, και χρειάστηκε να πάρω και προσωπικό κόστος, όπως ε, ε, και πολλές άλλες γυναίκες και στην Κροατία και στην Ευρώπη. Έχουμε αγωνιστεί ως γυναίκες για πολύ για να εξασφαλίσουμε την ισότητά μας και ο αγώνας μας συνεχίζεται. Υπάρχουν δηλαδή προσπάθειες και επιτεύγματα που θα πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά. Δηλαδή έχουμε κάνει θαύματα αλλά δεν έχουμε φτάσει εκεί που πρέπει σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή εάν δούμε μια μεγάλη συνέλευση ενός διεθνούς οργάνου, για παράδειγμα ε, τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, τον ΟΑΣΕ ή το Συμβούλιο της Ευρώπης, θα διαπιστώσετε ότι οι γυναίκες αποτελούν την μειοψηφία. Αλλά αυτό ισχύει και εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και στα Εθνικά Κοινοβούλια των περισσότερων κρατών μελών παρότι ο αριθμός ε, των γυναικών ε, σε όλα αυτά τα όργανα έχει αυξηθεί κατά τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, θα πρέπει να κάνουμε περισσότερο. Όλοι μας θα πρέπει να επιτύχουμε περισσότερα. Η Ευρώπη θα πρέπει να συνεχίσει να έχει τον ηγετικό εδώ ρόλο και να χαράσει την πορεία για ολόκληρο τον κόσμο. Βλέπουμε λοιπόν να υπάρχουν και σε αυτόν τον αιώνα ακροτηριασμός των, ε, γενετικών οργάνων, εμπορία ανθρώπων, άρνηση σε ό,τι αφορά το δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην πρόσβαση στην δημόσια υγεία, ε, το δικαίωμα επιλογών για τις γυναίκες. Βλέπουμε ε, βία, βλέπουμε σειράξεις, βλέπουμε τρομοκρατία. Και φυσικά όλα αυτά τα προβλήματα δεν επηρεάζουν μόνο ε, ναρακορίσια και γυναίκες, αλλά και τους άνδρες και τα αγόρια, αλλά ε, συχνά οι γυναίκε είναι εκείνε που είναι κύριοι διαμεσολαβητές και για την ειρήνη. Η διαμεσολάβησή τους είναι ε, απολύτω απαραίτητη για την χρηστή διακυβέρνηση, για τη δημοκρατία και έχει ε, αποδειχθεί επί τη βάση στατιστικών ότι όταν οι γυναίκε συμπεριλαμβάνονται στι διαδικασίε συμφιλίωση και ανοικοδόμηση, οι εν λόγω διαδικασίε έχουν πολύ περισσότερε πιθανότητε επιτυχίε. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε πολύ περισσότερε γυναίκε στου μηχανισμού πρόληψη και επίλυση διαφορών και γενικότερα υψηλότερη συμμετοχή του στην πολιτική ζωή. Κατά τι επιθέσει που δέχτηκε η Κροατία, οι γυναίκε μα ε, υπερασπίστηκαν τη χώρα μα ε, πλευρό πλευρό με τους, ε, με τους άντρες ε, και εργάστηκαν σε μία σειρά αποτομίας ε, και έπαιξαν ηγετικό ρόλο και μετά από τη σύγκρουση, στο πλαίσιο δηλαδή της αποκατάστασης και της ανοικοδόμησης. Άρα λοιπόν ο ρόλος της γυναίκα, γυναίκας στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών είναι αναντικατάστατος. Αν τους δοθούν οι κατάλληλοι πόροι και οι κατάλληλες δυνατότητες και εφόσον περιλαμβάνονται στις βασικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων μπορούν να αποτελέσουν πραγματικά ηγετικό να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε αυτέ τι διαδικασίε. Χωρί αυτέ, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η ειρήνη. Εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων παίζει καθοριστικό ρόλο για όλου ε, τους γνωστούς λόγους. Αλλά σε ό,τι αφορά του σκεπτικιστέ και εκείνους που επιμένουν να μα αμφιβάλλουν, ε, θα του αναφέρω ένα πολύ πιστικό επιχείρημα, την οικονομία δηλαδή. Ε, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι ε, Στι ε, οικονομίε εκείνε όπου έχουμε περισσότερες γυναίκε και σε διευθυντικέ και μη θέσει, η οικονομία αυξάνεται ταχύτερα, το ΑΕΠ ε, έχει μεγαλύτερου ρυθμού αύξηση, περισσότερη απασχόληση ε, και καλύτερη αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται από τη γύραση του πληθυσμού. Η αύξηση τη ισότητα μεταξύ των δύο φύλων μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ κατά 6,1 έως 9,6%, γεγονός που αντιστοιχεί για την Ευρώπη σε 15 δισεκατομμύρια ευρώ και στις χώρες εκείνες όπου η δυνατότητα αυτή πραγματικά υφίσταται όπως στην Κροατία, το δυναμικό για αύξηση του ΑΕΠ φτάνει έως και το 12%. Υπάρχουν λοιπόν οικονομικά ωφέλη και ε, στις ε, ε, κοινωνίες όπου υπάρχει πραγματικά οικονομική επιτυχία ισχύει το ότι δεν υπάρχουν αποκλεισμοί και οι γυναίκες συμμετέχουν στην εξουσία. Αντιθέτως στι ε, χώρε εκείνε όπου δεν υφίσταται κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει ελευθερία επιλογών για τι γυναίκε. Η οικονομική δηλαδή εξάρτηση και σε χώρε του αναπτυσσόμενου και του ε, ανεπτυγμένου κόσμου υπάρχουν ε, μία σειρά από προβλήματα που μπορούν να οδηγήσουν και στην ενδοοικογενειακή βία. Και η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη ε, στις ε, χώρες εκείνες όπου οι γυναίκες ε, τη χάνουν χειρότερες μεταχείρισεις από ό,τι και κατοικίδια ζώα. Και δυστυχώς έχω βιώσει, έχω υπάρξει μάρτυρα τέτοιων καταστάσεων. σε ό,τι αφορά την ενδοοικογενειακή βία θα πρέπει να πω ότι τα δικαστήρια ακόμα και στην Κροατία δεν είναι αρκούντες αυστηρά με εκείνου που προβούν σε αυτά τα αδικήμενα. Και ε, συχνά, για παράδειγμα, σε εγκλήματα σεξουαλική βία, αυτά αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό από τα δικαστήρια. Και α μην ξεχνάμε το βιασμό που χρησιμοποιείται ως όπλο στο πλαίσιο, της, ε, στο πλαίσιο σειράξεων και πολέμου. Συχνά στον, ε, στην απασχόληση έχουμε χαμηλότερους μισθούς για τις γυναίκες, υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας ε, αντιμετωπίζει περισσότερα προβλήματα ε, λόγω της ε, δημιουργίας οικογένειας αργότερα. Δηλαδή αντιμετωπίζονται με δυσπιστία σε ό,τι αφορά την ε, εξέβρεση εργασία Ωστόσο έχουμε γυναίκες παντού, επιστήμονες από πυρηνικές φυσικούς μέχρι και πολιτικούς. Και ταυτόχρονα αυτές οι γυναίκες είναι μητέρες, είναι σύζυγοι. Και συχνά αναγκάζονται να εργάζονται πολύ περισσότερο από ότι οι άντρε για να καταφέρουν να επιτύχουν. Και αυτό αποτελεί μια μεγάλη επιβάρυνση για μα. Παρ' όλα αυτά, προσπαθούμε συνέχεια και αποδεικνύουμε κάθε μέρα ότι είμαστε σε θέση να τα καταφέρουμε. Και όχι απλά τα καταφέρνουμε, πραγματικά ε, επιτυχάνουμε αριστεία Και γι' αυτόν ε, το λόγο είμαστε ακριβώς ε, ε, στον ίδιο βαθμό ικανέ ε, και έχουμε τα ίδια προσόντα όπω και οι άντρε για να συμμετέχουμε στι όλε διαδικασίε και στι ε, πολιτικέ και ίσω είμαστε ακόμα και καλύτερε από του άντρε. Ωστόσο, έχω διαπιστώσει, για παράδειγμα, πω όταν, για παράδειγμα, οι πρωθυπουργοί εξετάζουν τους, ε, ποιου θα επιλέξουν ω υπουργού, εξετάζουν κυρίω άντρε και μετά τι κάνουν, λένε Α, θα πρέπει δυστυχώ να συμπεριλάβω και κάποιε γυναίκε μέσα στη σύνθεση των υπουργών. Ε, δυστυχώ αυτή είναι η διαδικασία και οι ποσοστό που ισχύουν για τι γυναίκε ε, συχνά δεν την χάνουν σεβασμό ε, σε διάφορε χώρε. Δηλαδή το ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται στι σχετικέ λίστε. Και ε, γυναίκε στον ε, παρτιάρισμό. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια γενική αλλαγή τη νοοτροπία, τη συλλογιστική μα. Θα πρέπει δηλαδή να καλλιεργήσουμε μια πολιτική κουλτούρα η οποία θα ευνοεί την ίση συμμετοχή στα κοινά των γυναικών. Θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα φιλοδοξία στις, ε, στα νεαρά κορίτσια μας. Ας τους πούμε τι μπορούν να κάνουν και τι δεν μπορούν να κάνουν. Ας μην διαχωρίζουμε τον κοινωνικό ρόλο ανδρών και γυναικών. Από εμά εξαρτάται δηλαδή να αλλάξουμε τα στερεότυπα σε ό,τι αφορά τα φύλλα που συνεχίζουν να ισχύουν ε, μέχρι και σήμερα. Αρνούμε να ε, δεχτώ ε, τα επιχειρήματα σε σχέση με την κουλτούρα που αναφέρονται σε σχέση με τις γυναίκες. Δεν υπάρχει δηλαδή κουλτούρα η οποία επιτρέπεται να εισάγει διακρίσεις βάρος γυναικών σε σύγκριση με τους άντρες. Η πολιτιστική κληρονομιά λοιπόν και τα ήθη και τα έθιμα, τα πολιτισμικά, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως απολογία για τη μη ανάληψη δράση ε, σε περίπτωση όπου υπάρχουν ε, δικαιώματα των γυναικών στην εναφιβόλου και σε ό,τι αφορά ε, μετανάστε, θα πρέπει και εδώ να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι αφορά την κατάσταση των γυναικών. Τα στερεότυπα δεν αποτελούν δηλαδή μέρο μια κουλτούρα ή μια θρησκεία. Όχι, θα πρέπει να τα αφαιρέσουμε από, το, από τη σχολική ύλη, από τα μέσα ενημέρωση, γενικότερα από την κοινωνική ζωή. Θα πρέπει δηλαδή επιτέλου να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τέτοιου είδου επιχειρήματα. Θα πρέπει να προωθήσουμε τον ρόλο των ε, γυναικών ε, και να επιτρέψουμε στι γυναίκε αλλά και στου άνδρε να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια. Για να το επιτέχουμε λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι ε, σημαντική ακριβώς για να επιτρέψει αυτή την αλλαγή της νοοτροπίας ε, και να ε, δώσει τις δυνατότητες για ένα καλύτερο μέλλον για τι γυναίκε και γενικά για την ανθρωπότητα. Χρειαζόμαστε λοιπόν διαδικασίε χωρίς αποκλεισμού χρειαζόμαστε ίσες ευκαιρίες και κανένα δεν θα πρέπει να διχάνει τι μενέστερε μεταχείριση. Θα πρέπει να συμμετέχουν ε, γυναίκε σε όλα τα ε, αναπτυξιακά προγράμματα και να λαμβάνεται αυτή η πτυχή υπόψη γιατί αυτό είναι το καλύτερο εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μα για να επιτύχουμε ισότητα των φύλων. Κυρίε και κύριοι, ο ρόλο των μέσων ενημέρωση είναι καθοριστικό. Δηλαδή θα πρέπει να εκπροσωπούν με ισόρροπο τρόπο γυναίκες και άντρες. Οι γυναίκες στην πολιτική έχουν χρειάζεται να υπομείνουν πολλά και εγώ δεν αποτελώ εξαίρεση, αλλά έχω μάθει να το αντιμετωπίζω και να συνεχίζω να επιμένω έτσι ώστε ο κόσμος μας να γίνει πιο φιλικός για τις κόρες μας. Εκείνοι που είναι αντίθετοι στις ε, ε, θέσεις μας θα κάνουν ό,τι μπορούν για να ε, κριτικάρουν τον τρόπο με τον οποίο δίνεστε, τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεστε, την κόμωσή σας, οτιδήποτε άλλο. Θα προσπαθήσουν να σας αποθαρρύνουν, θα προσπαθήσουν να σας ασκήσουν κριτική και θα προσπαθήσουν να επιβάλλουν σε εσά κανόνε οι οποίε υποτίθεται πω ισχύουν μόνο για τι γυναίκε. Αλλά όλοι αυτοί ε, το κάνουν ακριβώ επειδή δεν ξέρουν ε, κάτι καλύτερο. Ε, και συνήθως επειδή φοβούνται, φοβούνται το δυναμικό το δικό μας ως ε, γυναικών. Οπότε το μήνυμα που έχω να περάσω σε όλα τα κορίτσια και τις γυναίκες είναι ε, να έχετε πίστη και να είστε εμπισμένες για τις ε, δυνατότητές σας, τις γνώσεις σας, τις δεξιότητές σας, τις ικανότητές σας και υπερασπιστείτε τον εαυτό σας. Είμαστε όλο ένα και περισσότερο τη σήμερα ημέρα και γυναίκες και άντρες που θα σας υποστηρίξουμε σε αυτή την προσπάθεια και με την αποφασιστικότητα που θα επιδείξετε θα καταφέρουμε να υπερκεράσουμε όλα τα εμπόδια που παραμένουν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Τώρα είναι μεγάλη μου χαρά που μπορώ να απευθύνω το καλώς ορίσατε στην Επίτροπο Γιούροβα που είναι υπεύθυνη για το χαρτοφυλάκιο καταναλωτών και ισότητας φύλων και ασφαλώς είναι από τους ισχυρότερου εταίρους μας και υποστηρικτές στον κοινό μας αγώνα υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φίλων. Κυρία Πίτροπε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμες και αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε σήμερα στη σημερινή σας δηλαδή συνεδρίαση. Θα αρχίσω με μια κάπως συναισθηματική νότα Φοβούμαι ότι είναι και η τελευταία ευκαιρία που θα έχω για να συμμετάσχω σε αυτό το παραδοσιακό, σε αυτή την παραδοσιακή εκδήλωση που σχετίζεται με την επέτειο της, ε, με την εορτή των γυναικών δηλαδή, ως επίτροπος. Θα αρχίσω λοιπόν πρώτα με την έκφραση ευχαριστειών προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την θαυμάσια συνεργασία που είχαμε έως τώρα. Ούτε μπορώ πια να υπολογίσω, να μετρήσω πόσες κοινοβουλευτικέ ερωτήσεις έχω λάβει, πόσες ώρες έχω περάσει στη μεγάλη αίθουσα του ημικυκλίου του Κοινοβουλίου, είτε στο Στρασβούργο είτε εδώ, πόσες φορές έχω ακούσει από την κυρία Πρόεδρο, από την κυρία Γκαρσία Πέρες, από άλλες ευρωβουλευτέ που τις βλέπω να κάθονται εδώ, να μου λένε «Γιούροβα, πρέπει να κάνει ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια». Ταυτόχρονα, άκουγα από το κοινοβούλιο ότι ζητούσε περισσότερα ταυτόχρονα όμως μου έλεγε δεν, είναι, δεν είσαι μόνη σου, θα σε βοηθήσουμε. Και νομίζω ότι επιτύχαμε κάποια πράγματα. Έχετε στο φυλάδιο που σας δείχνω τους νέους αριθμούς. Ακόμα το πιάνουν ζεστό το εντυπώ διότι βγήκε μόλις από το τυπογραφείο. Προσοχή λοιπόν μην κάψετε τα δαχτυλά σας. Βλέπετε εδώ δεδομένα που δείχνουν κάποια πρόοδο. Όμως ταυτόχρονα δείχνουν τα νούμερα αυτά ότι μένουν πολλά πράγματα ακόμη να γίνουν. Και γι' αυτό το λόγο εγώ ειδοποίησα τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα μιλώντας προσωπικά με τους ε, ηγέτες τους για να προβάλλουν όσο το δυνατόν περισσότερες γυναικείες υποψηφιότητες στα ψηφοδέλτια, διότι η δουλειά μας αυτή πρέπει να συνεχιστεί. Και μια φράση ακόμη για τον αγώνα αυτό. Στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας έλαβα πολλές ερωτήσεις και από πολλούς άνδρες με πολύ ισχυρή κινητοποίηση. Δεν είναι μόνο οι γυναίκες δηλαδή που ενδιαφέρονται για το θέμα. Το πρόβλημα ότι δεν έχουμε αρκετές γυναίκες σε θέσεις που λαμβάνουν αποφάσεις και ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Αυτό δεν το κάνουμε μόνο για να εξυπηρετήσουμε τις γυναίκες, δεν αποτελεί προνόμιο, είναι υποχρέωση. Ακόμα ε, θεωρείται κάπως ως προνόμιο ε, υπέρ των γυναικών, όμως κυρίες και κύριοι, εδώ είναι το πρόβλημα κοινωνικό. Διότι υπάρχει κάτι το μη υγιές στην κοινωνία μας. Άνω το 60% των γυναικών έχουν πτυχία πανεπιστημίου και κάπου εξαφανίζονται. Ωστόσο, θα σας δώσω και άλλα δεδομένα τέτοια, αλλά πριν να προχωρήσω σε αυτό θα ήθελα να σας αναφέρω κάποιες παρατηρήσεις. Ποιο είναι αυτό το πράγμα που δεν είναι υγιές. Ε, έχουμε τόσες ευθύνε ως γυναίκες, αλλά δεν έχουμε εξισορρόπηση όσον αφορά την εξουσία που ασκούμε. Υπάρχει λοιπόν κάπου ένα συστημικό λάθος. Τα λέω με κάπως τεχνικό τρόπο, αλλά αν δείτε τα νούμερα θα το δείτε αυτό καθαρά βλέπετε ότι με αυτό το 60% των πτυχιούχων έχουμε 6% Chief Executive Officers, δηλαδή επικεφαλής επιχειρήσεων, σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Έχουμε ακόμα μεγάλο κενό στην απασχόληση. Είχαμε πει να φτάσουμε στο 75%, δηλαδή να είναι το ίδιο με τους άνδρες. Έχουμε περίπου 20% κατά μεσονόρο... όρο σε εισηγμένες επιχειρήσεις, στα συμβούλια εισηγμένων επιχειρήσεων. 30% γυναίκες βουλευτές στα εθνικά κοινοβούλια. 36,5% μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, ευρωβουλευτές δηλαδή. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά αλλάζει αυτό. Όμως κάπου κάπου ακόμη κάποιε κυβερνήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν καθόλου γυναίκες στους κόλπους τους. Αν κατέβουν κάποια στιγμή οι Αριανοί εδώ στην γη και δουν αυτά τα πράγματα, δεν θα έχουν καμιά κατανόηση. Μιλώντας στατιστικά είπα εγώ ότι εργάζομαι υπέρ των μειονοτήτων που είναι οι άνδρες δεν θα, δεν θα κατονομάσω τις κυβερνήσεις αυτές που δεν έχουν καθόλου γυναίκε υπουργού. Κάτι τέτοιο όμω ωστόσο είναι πολύ μειοπικό και ε, καθόλου σόφρον. Άρα έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχαμε τον στόχο 40% γυναίκες σε ανώτερες διοικητικές θέσεις. Κοντεύουμε να το φτάσουμε το ποσοστό αυτό. Έχουμε λίγο πάνω από 39%. Πηγαίνει σιγά σιγά, αλλά πηγαίνει καλά. Αλλά δεν είναι και αυτόματο αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε κάποια ποσόστοση και εκεί οι άντρες ίσως αισθάνονται ότι εξαπατούνται. Είναι απολύτως έντιμος ο ανταγωνισμός. Ίσως δεν χρειάζονται καν θετικά μέτρα υπέρ των γυναικών δηλαδή. Αρκεί ο έντιμος ανταγωνισμός, διότι υπάρχουν γυναίκες οι οποίες ε, ε, έχουν και ε, τον ενθουσιασμό και τα προσόντα για να καλύψουν τις σχετικές θέσεις. Και θεωρούμε ότι πρέπει όντως να προετοιμάζονται οι γυναίκες για τις θέσεις αυτές. Κάνουμε σεμινάρια, εκπαιδεύσεις, έχουμε ένα είδος mentoring, έχουμε διαδικτύωση. Όλα αυτά τα πράγματα όμως είναι αποτέλεσμα προσπάθειας, δεν γίνονται αυτομάτως. Αποδίδουν όμως. Επανέρχομαι στις χώρες μέλη. Η Ισπανική κυβέρνηση τώρα έχει πλειοψηφία γυναικών. Έτσι δεν είναι. Υπάρχει ποσόστοση. Κυρία Γκαρσία Πέρες, τι λέτε, βλέπετε ότι επαγρυπνεί η κυρία Γκαρσία Πέρες. Νομίζω ότι η συμμετοχή των γυναικών έχει φτάσει στο 67% στην κυβέρνηση. Λοιπόν, Έχουμε Υπουργό Οικονομίας, ε, Υπουργό Οικονομικών, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης σημαντικές θέσεις, σημαντικά χαρτοφυλάκια που παλιά ήταν, τα είχαν οι άντρες. Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενημερωτική αυτή ε, παρέμβασή σας. Ακούν καμιά φορά άντρε αυτά που λέω, ζητούμε περισσότερε γυναίκε, περισσότεροι εξουσιαστέ γυναίκε, διότι ούτω ή άλλω αναλαμβάνουν πάρα πολλέ ευθύνε. Ακούω καμιά φορά τι φωνέ να λένε Α, ζητάτε καυγά. Ζητάτε να μας αντικαταστήσετε. Και αυτό που λέω εγώ είναι όχι. Θέλουμε να εξισορροπήσουμε, να εξισορροπήσουμε μάλλον ευθύνε με εξουσία. Και θέλουμε να συνεργαστούμε. Διότι οι γυναίκε παίζουν πολύ καλά <clears throat> όταν παίζουν σε ομάδα. Θέλουμε συνεργασία λοιπόν, αλλά με έντιμους όρους, να πάλι αυτή η λέξη fairness, δίκαιοι όροι, έντιμοι όροι, όταν είναι ιδιαίτερα εχθρική η ατμόσφαιρα, λέω, κοιτάξτε, δεν θέλουμε καυγάδε. Μα αρέσει για μια φορά, σας αγαπάμε κιόλα. Λέω στου άνδρε, δηλαδή, συνομιλητέ μου. Αυτή είναι η θέση μου. Δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε του άνδρε, ούτε θέλουμε να μαλώνουμε μαζί του. Τώρα κάπω πιο σοβαρά. Η κυρία Πρόεδρο μίλησε για την βία και τα απαράδεκτα αυτά φαινόμενα στην κοινωνία μας. Εμείς ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να μπουν στην πολιτική, στις μεγάλες επιχειρήσεις, σε θέσεις ε, διοικήσεων επιχειρήσεων, ε, να αρχίσουν να συμμετέχουν σε θέσεις που είναι ανοιχτές και ορατές στην κοινωνία. Όλο και, περισσότερο, όλο και περισσότερες γυναίκες ε, απειλούνται ωστόσο διαδικτυακά. Απειλείται η σωματική τους ασφάλεια. Υπάρχει πολλή παρενόχληση και απειλή βίας και κατά γυναικών ευρωβουλευτών και υποψηφίων και πρόκειται για κάτι που μας ανισχύει και περισσότερο. Είναι όμως ένας αποθαρρυντικός παράγων, αυτός που ακούω από νέες, νεαρές γυναίκες, τις οποίες καλό να προσέλθουν στην πολιτική, αλλά και από γυναίκες δημοσιογράφους, που λένε αντιμετωπίζουμε φοβερές επιθέσεις διαδικτυακής απειλής και βίας. Τόσο πολύ που σκεπτόμαστε να κάνουμε κάτι άλλο καλύτερα για να έχουμε εγγυημένη την ασφάλεια τη δική μα και την ασφάλεια των οικογενειών μα. Πρόκειται για μια τάση η οποία πρέπει να σταματήσει. Ε, θέλω από πολύ καιρό να μιλήσω για το πράγμα αυτό. Πολύ συχνά έρχομαι σε επαφή με αυτόν ε, τον τομέα της ηλεκτρονικής τεχνολογίας πληροφορικής, αλλά πρόκειται για μια απειλή και μια βία που όχι μόνο είναι απαράδεκτη, αλλά και είναι και παράνομη. Ε, διώκεται από τον νόμο, από κάθε άποψη. Η κυρία Πρόεδρος μίλησε για την βία κατά των γυναικών αλλά και κατά παιδιών. Για την οικιακή βία έχουμε συγκλονιστικά νούμερα. Μία από μία σε τρεις γυναίκες άνω των 15 έχει νιώσει, έχει ε, υποστεί κάποιο είδους βία λέω ότι στην Ευρώπη είναι ασφαλή οι γυναίκε, αλλά όταν βλέπω τα νούμερα αυτά, για μένα ξαναλέω είναι συγκλονιστικά και απολύτω απαράδεκτα. Και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε εργαλείο που διαθέτουμε ω πολιτική και στο επίπεδο των χωρών μελών και στο ευρωπαϊκό. Δηλαδή, νομοθεσία. Επομένω, εδώ μιλώ για το ποινικό δίκαιο. Πρέπει να το εξετάσουμε αυτό το ενδεχόμενο. Καλύτερε εκστρατείε, χρηματοδότηση, εκπαίδευση των επαγγελματιών επιβολής του νόμου για ε, τη διεξαγωγή εκστρατιών. Γνωρίζετε ήδη από το 2017 υπάρχει μια διαρκή εκστρατεία κατά τη της κατά της βίας, κατά των γυναικών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί, γιατί μέρος της κοινωνίας μας θεωρεί ακόμη ότι η βία είναι κάτι το αναπόφευκτο. Είναι φυσιολογικό. Και πιθανότατα το θύμα της βίας το προκάλεσε την προκάλεσε την βία αυτή. Δηλαδή επικαλούνται αντικειμενικούς λόγους που δικαιολογούν υποτίθεται τη συμπεριφορά του δράστη. Αυτή είναι η εικόνα που έχει συχνά η κοινωνία μας. Και απέναντι σε αυτήν πρέπει να αγωνιστούμε. Ακούσαμε άλλωστε από την κυρία Πρόεδρο της, της ε, ε, Κροατίας, με ενέπνευσε πραγματικά, ότι οι πολιτισμικές παραδόσεις δεν μπορούν να αποτελούν ε, δικαιολογίες στην περίπτωση αυτή, όχι μόνο στην περίπτωση της βίας. Έχουμε άλλωστε στατιστικές που δείχνουν ότι περίπου μισό εκατομμύριο νεαρές γυναίκες και νεαρά κορίτσια υφίστανται αυτόν τον, τον βάρβαρο ακροτηριασμό των γεννητικών οργάνων. Και όταν μιλώ καμιά φορά με ανθρώπους που εργάζονται στις δυνάμεις ασφαλείας, λένε «Α, κοιτάξτε, είναι μέρος της πολιτιστικής παράδοσης αυτών των ανθρώπων». Μου έρχεται να τους σκοτώσω τότε. Διότι είναι απολύτως απαράδεκτο αυτό. Πρέπει να διωχθεί, πρέπει να εξηγηθεί στην κοινωνία ότι ο κάθε ένας και κάθε μία έχουν το καθήκον να καταγγείλουν ότι κάτι τέτοιο πάει να γίνει. Δηλαδή ότι γίνονται προετοιμασίες για να γίνει αυτός ο τελετουργικός ακροτηριασμός εν τέλει. Αυτές οι πολιτισμικές προφάσεις είναι ανεπίτρεπτες για ολόκληρη την κοινωνία και για τα πρόσωπα τα οποία τώρα έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οφείλουμε να έχουμε ένα πάρα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ευρωπαία γυναίκα είναι ατομικά ελεύθερη και ισχυρή και έχει το δικαίωμα να αποφασίσει μόνη της η ίδια αν θα σπουδάσει, αν θα εργαστεί και πού θα εργαστεί, αν θα παντρευτεί, πόσα παιδιά θα κάνει, αν θέλει να κάνει. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά, αυτά, αυτές είναι οι ιδιότητες της Ευρωπαίας γυναίκας και πρέπει να είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι και να αγωνιζόμαστε για την ισότητα των φίλων, διότι αν όχι, το λέω και το ξαναλέω, θα είμαστε μόνο υποκριτές. Δηλαδή θα μιλούμε χωρίς τα λόγια μας να τα ακολουθούν έργα. Όταν κάθομαι εδώ είμαι και κάπως, ε, ε, είμαι και περισσότερο παθιασμένη όταν τα λέω αυτά τα πράγματα. Έχω ε, τη συνέστηση ότι μακρηγορώ, αλλά Τελειώνω τώρα. σω μου χρειάζεται ένα λεπτό ακόμη, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, έρχονται οι εκλογές. Χάρη στο γεγονός ότι έχω περάσει πολλές ώρες στην Ολομελιά σας, γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι μετά την 26η Μαΐου να υπάρχουν υπεύθυνοι και ευφύ άνθρωποι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μια, ένα καλό μείγμα εθνών, παραδόσεων, γυναικών ανδρών, νέων, πρεσβύτερων, μια καλή ισορροπία καλών ανθρώπων. Αυτό χρειάζεται η Ευρώπη, αυτό χρειαζόμαστε όλες και όλοι μας. Και αυτή είναι η ευχή μου. Και ενθαρρύνω τις γυναίκες να προχωρήσουν και να προβάλλουν υποψηφιότητες. ευχαριστούμε, Επίτροπε. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Βιργινία Λάγκμπακ, Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων. Θα μας παρουσιάσει μια πλήρη εικόνα για την παρουσία των γυναικών στην πολιτική σήμερα. Κυρία Λάγκμπακ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είδα ότι οι ομιλητές σας έδωσαν ήδη επιχειρήματα και εγώ θα σταθώ σε αυτά, αλλά με νούμερα για να σας ε, αποδείξω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε, να δουλεύουμε, να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας. Ας ξεκινήσω από κάποια από τα στοιχεία που συζητήσαμε τους δημοσιογράφους πριν λίγες μέρες και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων τα γνωρίζουν. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα είναι ότι αν δούμε, αν σταθούμε στη χρονιά του 1979 που για πρώτη φορά εξελέγει με απευθείας εκλογές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είχαμε 17% γυναίκες. 40 χρόνια μετά έχουμε κάτι παραπάνω από τα διπλάσια, το διπλάσιο ποσοστό δηλαδή. Γιατί η πρόοδο είναι τόσο αργή. Ας το σκεφτούμε λιγάκι. Έχουμε τον δείκτη για την ισότητα των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αν είχαμε, ήμασταν στο 100, θα ήμασταν ίσοι, άντρες και γυναίκες. Βλέπουμε πόσο μακριά είμαστε, πόσο απέχουμε. Είμαστε λίγο πιο κάτω από το 50. Και βλέπετε μάλιστα με βάση το δίχτυ που βρίσκεται η χώρα σας. Για την, στην πολιτική εξουσία, στην οικονομία. Βλέπετε που είναι οι γυναίκες ε, σε θέσεις σημαντικές. Το κενό είναι πολύ μεγάλο γενικά. Και όπως είπε η Επίτροπος, αυτό συμβαίνει τον 21ο αιώνα. Όταν κοιτάτε αυτά τα νούμερα, ρωτάστε ποια είναι τα αίτια. Ας πούμε, τα μέλη του, του Κοινοβουλίου, κατά μέσο όρο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, έχουμε ένα ποσοστό. Στα Εθνικά Κοινοβούλια τα ποσοστά αυτά είναι χαμηλότερα. Ε, για τους υπουργούς, υπουργικές θέσεις, γυναίκες στο Κοινοβούλιο είναι περίπου ίδιες. Επίσης, έχουμε ένα εργαλείο που φτιάξαμε πέρυσι για να δούμε για ποιο λόγο οι γυναίκες δεν μπορούν να ανέλθουν. Ε, αναλύουμε και την κουλτούρα και την οτροπία, ε, πι, πιθανότητες παρανόχλησης, όλες τις τροχοπέδες ε, που παρεμποδίζουν τις γυναίκες να φτάσουν σε ηγετικέ θέσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από ό,τι ξέρω, και ο Γενικός ε, Διευθυντή για την Ανάπτυξη αναπτύσσουν κάποια εργαλεία για να δούμε πώς θα στηρίξουμε τις γυναίκες, όπως μια εκτίμηση από ομότιμους ε, και κάποιες καλές πρακτικές. Φυσικά η Επίτροπος θα μπορούσε να σας πει περισσότερα, αλλά προσπαθούμε να καταλάβουμε τους λόγους και τους λανθάνοντες ακόμα λόγους που δεν, τους, δεν έρχονται εύκολα στο μυαλό ε, για να καταλάβουμε και να αναλύσουμε τα φαινόμενα αυτά. Επίσης ε, ακούστηκε η λέξη ποσοστώσεις. Δεν θέλω να το συζητήσουμε πολύ, αλλά το αναλύσαμε το θέμα και βρήκαμε ότι η ποσόστοση δεν είναι η εξήγηση ή δεν είναι το φάρμακο, δεν είναι πανάκια. Είναι ένας από τους τρόπους για να ξεκινήσει η αλλαγή. Τον Οκτώβριο του 19 θα έχουμε το νέο δίχτυ για την ισότητα των φύλων και βλέπουμε ότι αυτά τα νέα κράτη-μέλη που έχουν ποσοστώσεις, ε, από αυτά τα 9 τα 8 έχουν καταφέρει να αυξήσουν τη συμμετοχή των γυναικών στην εξουσία, σε θέση εξουσίας, εκτός από την Κροατία. Άρα η ποσόστοση είναι ένα ενδιάμεσο μέσο. Μας κάνει να σκεφτόμαστε η πρόεδρο μα είπε ότι τα κόμματα σκέφτονται καταρχήν του άντρε και μετά στο τέλο βάζουν και κάποιε γυναίκε. Αλλά χάρη ποσοστό, ίσω αλλάζουν κάποια πράγματα. Τι συμβαίνει λοιπόν. Κάναμε μία μελέτη εξ ονόματος της Αυστριακής ε, Προεδρίας, όπου είδαμε ότι τα νέα κορίτσια είναι πολύ εκτεθειμένα στο, στην παρενόχληση και στο διαδίκτυο, ε, λόγω της τάσης, ε, λόγω της έλλειψης ε, ανοχής που υπάρχει από το κοινό, δεν δέχεται ο κόσμος να μιλάνε με τον τρόπο που μιλάνε. Δεν δεχόμαστε αυτό να είναι, δεν το δεχόμαστε, δεν είναι επιτρεπτό και δεν δεχόμαστε το πολιτιστικό επιχείρημα. Δέκα χώρες συμμετείχαν σε μία έρευνα ε, και ρωτήσαμε διάφορα κορίτσια και γυναίκες, νεαρές γυναίκες, για να μας πούν για ποιο λόγο δεν θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική. Και είδαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές ε, στο πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Πέρασαν 40 χρόνια, κινούμαστε με το ρυθμό της χελώνας, είναι απαράδεκτο αυτό Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες προτάσεις και εκστρατείες, ε, συμμετέχουν και πολλές ΜΚΟ. Πολλές ε, οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών ασχολούνται με αυτό το θέμα της ότας των φύλων. Πρέπει να προχωρήσουμε, πρέπει να επιταχύνουμε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Πρέπει να αλλοϊποστηριχθούμε, οι γυναίκες να στηρίξουν τις γυναίκες και οι άντρες να υποστηρίξουν επίσης τις γυναίκες. Ελπίζω ότι εν ώψη των εκλογών πολλές γυναίκες θα ψηφίσουν θα σταυρώσουν γυναίκες, αλλά και πολύ περισσότερες γυναίκες θα συμμετάσχουν στην πολιτική. Ευχαριστώ για την ε, ομιλία σας αυτή. Και τώρα θα παραδώσω τη σκητάλη του Προέδρου. Θα δώσω το λόγο στους δύο ε, Προέδρους των πάνελ που θα συζητήσουν την πραγματική εξουσία των γυναικών στην πολιτική και πώς θα την τονώσουμε και την ε, συμμετοχή των νεαρών γυναικών στην πολιτική. Θα ήθελα το πρώτο πάνελ, οι ομιλητές του πρώτου πάνελ να έρθουν εδώ στο βήμα. Η κυρία Γνιέσκα Κοσλόσκα Ράζινιτς από την Πολωνία και που, ήταν ε, πρόεδρος του, του, θα είναι πρόεδρος του πρώτου πάνελ, η κυρία Χενρίκα Μπόσνιατς, πρόεδρος της Πολωνικής Συνομοσπονδίας Λεβιάταν, αντιπρόεδρος του Business Europe και ιδρυτής του Συνεδρίου των Γυναικών από την Πολωνία. Η κυρία Μέριλ Κένι, λέκτορας για το, τα φύλλα και την πολιτική στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και η Ευρωβουλευτής Αγγέλικα Μλίνερ μέλος της Επιτροπής Γυναικών. Θα παραδώσω το, την Προεδρία του πρώτου πάνελ στην κυρία Αγνιέσκα Κοσλόφσκα Ράζιετς. γεια σας ε, σε όλους ε, και σας ζητώ συγγνώμη. Έτσι. Είμαι λίγο μπουκωμένη σήμερα, δεν έχω φωνή. Οπότε ίσως καλό είναι τώρα που θα έχετε και διερμηνία να ακούσετε τη διερμηνία γιατί είναι πιο ευχάριστη. Λοιπόν, ευχαριστώ ε, όλες ε, τις ε, ομιλήτριες μας σήμερα σε αυτό το πρώτο πάνελ σε σχέση με την πραγματική εξουσία των γυναικών στην πολιτική και το πώς μπορούμε να την ενθαρρύνουμε. Και καλωσορίζω στις τρεις ομιλήτριές μας την κυρία Ενρίκα Μπογνίαρ, την Μέριλ Κέρ και την Αγγέλικα Μλίναρ που συμμετέχει βέβαια ως μέλος εδώ της Επιτροπής ΕΦΕΜ. Προτού δώσω λοιπόν το λόγο σε αυτές τις εξαιρετικές ε, ομιλήτρες θα ήθελα να κάνω κάποια ε, εισαγωγικά σχόλια από τη δική μου πλευρά. Γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες ε, συμμετέχουν στην πολιτική ζωή και αυξάνονται οι αριθμοί αυτοί και τα ποσοστά της συμμετοχής τους στην πολιτική ζωή αλλά και σε υψηλές ε, θέσεις αλλά δεν επαρκούν όλα αυτά. Θα πρέπει δηλαδή να κάνουμε περαιτέρω προσπάθειες και θα πρέπει να συζητήσουμε τους λόγους οι οποίοι μας οδηγούν σε αυτήν την ε, τεράστια δυσαναλογία που βιώνουμε σήμερα σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση των γενικών στην ε, πολιτική. Ε, και βέβαια ε, εδώ έχουμε ε, να κάνουμε και με το ζήτημα γενικότερα της πρόσβασης στους απαραίτητους πόρους και, στις, και στον απαραίτητο χρόνο. Γιατί βέβαια όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους και στο πλαίσιο της, των προεκλογικών εκστρατιών. Και σε ό,τι αφορά ακριβώς αυτό το ζήτημα του διαθέσιμου χνώρου, ε, γνωρίζουμε ότι κάθε εβδομάδα οι γυναίκε κατά μέσο όρο εργάζονται 10 ώρε ε, περισσότερο και αυτό αντιστοιχεί σε 520 ημέρε ε, το χρόνο. Οπότε λάβετε υπόψη σα και προσπαθείτε να σκεφτείτε σε τι ακριβώ αντιστοιχούν 520 ώρε εργασία το χρόνο παραπάνω. Επίση, η πληροφόρηση αποτελεί κάτι το πολύ σημαντικό στον τομέα τη πολιτική, γιατί η πολιτική βέβαια ουσιαστικά έχει να κάνει με τον συμβασμό, με τη διαλλακτικότητα, όπου προσπαθούμε δηλαδή να συγχωνεύσουμε, αν θέλετε, διαφορετικέ και αντίθετε ιδέε. Άρα λοιπόν οι πληροφορίες εδώ ε, είναι πάρα πολύ σημαντικές και στο ίδιο πλαίσιο και η καταπολέμηση των στερεοτύπων με βάση τα οποία ε, ουσιαστικά ε, λαμβάνει η χώρα με υποτίμηση και μια παραγνώριση των δυνατοτήτων των γυναικών. Εγώ θυμάμαι πως μια συνάδελφος η οποία που ήταν 33 ετών είχε αναλάβει ως υπουργό ε, Αθλητισμού ε, ε, και οι δημοσιογράφοι ουσιαστικά προσπαθούν να αμφισβητήσουν και τις δεξιότητές της και την ηλικία της και αμφισβητούσαν το κατά πόσο ήταν έτοιμη για να αναλάβει αυτό το ρόλο. Ενώ άλλοι συνάδελφοι υπουργοί δεν έλαβαν τέτοιου είδους ερωτήματα επικριτικά. Απλώ ε, τα ερωτήματα που τέθηκαν από του δημοσιογράφου, εκείνου του άντρε υπουργού, ε, είχαν να κάνουν μόνο με τα ε, προβλήματα που ήθελαν να αντιμετωπίσουν, ποιες, ποια ήταν τα μέτρα που ήθελαν να λάβουν. Άρα λοιπόν το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι γιατί καλούνται συνέχεια οι γυναίκε να αποδείξουν κάτι σε κάποιον, γιατί θα πρέπει να, να αποδεικνύουν συνέχεια ότι είναι οι καλύτερε, οι εξέχουσε και ότι εργάζονται περισσότερο από του υπόλοιπου. Ένα ακόμα ε, φαινόμενο ε, που παρατηρείται είναι ουσιαστικά η παραγνώριση των γυναικών στην ε, πολιτική. Υπήρχε δηλαδή όταν εγώ εργαζόμουν στο Πολωνικό Κοινοβούλιο υπήρχε πραγματικά ένα ολόκληρο στρατό γυναικών οι οποίε εργάζονταν ω υφυπουργοί, γενικοί γραμματεί υπουργείων και μιλάμε δηλαδή για υψηλότατε θέσει Και ακριβώς επειδή δεν έχουν την ίδια, ε, την ίδια πολιτική ε, βαρύτητα με άλλες, ε, δεν υπήρχαν άντρες οι οποίοι προσπαθούσαν να τις καταλάβουν. Και είδαμε λοιπόν ότι όλες αυτές οι γυναίκες εργάζονταν πήρε το δός, ούτως ώστε να λάβουν βέβαια τα, τα ωφέλη και τη δόξα οι επικεφαλής τους, οι υπουργοί τους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο διαπιστώνουμε και ξανά και ξανά και στον τομέα της πολιτικής και σε άλλους τομείς. Και αυτό πραγματικά πραγματικά με εξοργίζει. Ε, και ε, απλώς και μόνο είναι αδικία. Δηλαδή, ε, μιλάμε για 40% που καταλαμβάνονται από γυναίκες αυτών των θέσεων, δηλαδή Υπουργών και Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, οι οποίε δεν αναλαμβάνουν υψηλότερε θέσει παρότι έχουν φτάσει τόσο ψηλά και θεωρούν δηλαδή ότι πραγματικά δεν έχουν καταφέρει αυτές οι γυναίκες να ε, λάβουν την απαραίτητη εξουσία. Ε, ε, δηλαδή παρότι ε, στα χαρτιά, αν θέλετε, ε, το αξίωμά του αυτό είναι υψηλό βαθμό, δεν έχουν πραγματική δυνατότητα και εξουσία για τη λήψη αποφάσεων. Άρα λοιπόν πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο για να τις ε, βοηθήσουμε, γιατί οι περισσότερε από εμάς δεν φτάνουμε ποτέ σε αυτές τις υψηλότατες θέσεις, σημαίνουμε πάντα στο παρασκήνιο. Άρα λοιπόν τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, σα καλώ όλε να συμμετάσχετε σε αυτήν την συζήτηση και ως πρώτη θα ήθελα να ζητήσω πρώτα από την κυρία Ενρίκα Μπόχνιαρτς να πάρει το λόγο η οποία κατάφερε να φτάσει πολύ ψηλά ε, και η οποία παραμένει σε τόσο υψηλή θέση. Εξηγήστε μας λοιπόν πώς μπορούμε να το επιτύχουμε. Παρακαλώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ η κυρία Μπόχνιαρτς. Δεν θα αναφερθώ στην ε, παρουσίασή μου, presentation δηλαδή. Αν τη θέλετε όμως, μπορείτε να μπορείτε να την ε, δείτε γιατί έχει μέσα πολλές πληροφορίες. Είχα την ευκαιρία και την τύχη να διαρευνήσω διάφορους κόσμους, και τον κόσμο της πολιτικής και τον κόσμο των επιχειρήσεων. Και εξετάζω τον ρόλο των γυναικών από τη σκοπιά της οικονομίας, γιατί είμαι και επαγγελματικά οικονομολόγος. Για μένα το πιο σημαντικό θέμα, και συζητούμε βέβαια για τον ρόλο των γυναικών εδώ τώρα και στην πολιτική αλλά και στις επιχειρήσεις. Το πιο σημαντικό λοιπόν για μένα είναι το γεγονός της απώλειας αυτής της ε, τεράστιας ε, δύναμης την οποία κρύβει μέσα της κάθε γυναίκα. Δεν είναι δυνατόν η κοινωνία να αφήνει να, σπαταλώνται, ε, να σπαταλάται αυτό το δυναμικό. Πρέπει να βρούμε τρόπους, μηχανισμούς που θα μας επιτρέψουν εν τέλει να επιταχύνουμε τη διαδικασία για να συμβάλλουν οι γυναίκες. Πρώτον, υπάρχει μεγάλη ομοιότητα ανάμεσα στον επιχειρηματικό κόσμο και στον πολιτικό κόσμο. Όταν η Αγνέσκα μίλησε για τον αριθμό υφυπουργών που έκαναν τη δουλειά του στην πολωνική κυβέρνηση, το ίδιο συμβαίνει στις επιχειρήσεις. Όταν πάτε σε μια μεσαία τράπεζα θα δείτε 80% των εργαζομένων είναι γυναίκες. 50% στη μεσαία ε, στο μεσαίο στρώμα των, ε, των, ε, των διοικητικών θέσεων. Τώρα, αν πάτε παραπάνω στα ανώτατα επίπεδα, θα δείτε ίσως μία γυναίκα. Το ίδιο σημαίνει στην πολιτική. Πρέπει να δούμε λοιπόν αυτούς τους δύο κόσμους, διότι και πάλι αλληλεξαρτώνται οι δύο αυτοί κόσμοι. Η Ανιέσκα μίλησε για το θέμα του χρήματος, που είναι σαφώς ένα από τα εργαλεία που ε, επιτρέπει έτσι τον αποκλεισμό των γυναικών από την πολιτική, διότι κανείς δεν μπορεί να υπάρξει στον κόσμο χωρίς χρήματα. Το πολύ σημαντικό για τις γυναίκες είναι η διαδικτύωση και πολύ περισσότερο από ό,τι για τους άνδρες. Διότι πρώτα-πρώτα Είμαστε εκεί για πολύ λιγότερο χρόνο και πρέπει λοιπόν να υπάρχει αλληλοκατανόηση μεταξύ των γυναικών. Έπειτα οι γυναίκε, αν θέλουν να κάνουν κάτι όλε μαζί, πρέπει να ε, συμπαθεί μεν, ε, ε, να συμπαθούν οι μεν τις δε. Αντίθετα με τους άντρες, γιατί εκεί τους άντρες ενδιαφέρει business μόνο. Δεν είναι ανάγκη να αλληλοσυμπαθιούνται. Από την άποψη λοιπόν αυτή θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία του συνεδρίου γυναικών που έχουμε φτιάξει και που έχει μια ζωή δεκαετών και που για πρώτη φορά δεν έχουμε την οργάνωση η οποία συγκεντρώνει τις γυναίκες στην πολιτική είτε στις επιχειρήσεις είτε στις μη, οργανώ... μη, ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ. έχουμε όλες μαζί. Και για 10 χρόνια ήταν πάρα πολύ σκληρή δουλειά αυτή που κάναμε για να αρχίσουμε να μιλούμε καν την ίδια γλώσσα. Διότι εγώ ως επιχειρηματίας για να μπορέσω να μιλήσω με την επικεφαλής του φεμινιστικού κινήματος στην Πολωνία ήταν σαν να μιλώ με άνθρωπο από άλλο πλανήτη και το ίδιο και με άλλους. Μετά από 10 χρόνια ωστόσο γνωρίζουμε πια ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει και τις γυναίκες στην πολιτική και τις γυναίκες στις επιχειρήσεις και τις ε, γυναίκες σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Νομίζω λοιπόν αυτή η λύση δεν ξέρω αν μπορεί να λειτουργήσει σε όλες τις χώρες, διότι για τέτοιου είδους οργάνωση δεν έχω ξανακούσει και είναι το πιο σημαντικό κοινωνικό κίνημα μετά από την αλληλεγγύη, τη Ολυνταρνόσκ στην Πολωνία το Κογκρέσο των Γυναικών. Αυτό που είναι επίσης πολύ σημαντικό ωστόσο είναι ότι έχουμε γυναίκες που κινητοποιούνται στις περιφέρειες και δεν σημαίνει δηλαδή ότι είναι μια ε, δομή με κάπως ηγετική μορφή και οι υπόλοιποι ας ακολουθήσουν. Υπάρχουν πολλές κινητοποιήσεις ε, από τα μικρά χωριά και τις μικρές πόλεις μέχρι, το, μέχρι ψηλότερα επίπεδα. Και στις τελευταίες τοπικές εκλογές λειτουργήσε καλά το σύστημα γιατί για πρώτη φορά είχαμε τον μεγαλύτερο αριθμό γυναικών που τελικώς αποφάσισαν να κατεβούν υποψήφιες. Από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα του Κογκρέσου των Γυναικών ήταν ότι το 2011 μπορέσαμε χρησιμοποιώντας αυτό το στενό παράθυρο ευκαιρίας που είχαμε τότε που κάπως ευνηδιάστηκε η πολιτική ζωή από το κίνημά μας μπορέσαμε να πάμε στην Βουλή και να πείσουμε τους βουλευτές, μιλώ πάντα για την ε, Δημοκρατία της Πολωνίας, να βάλουν ποσοστώσεις 35% γυναίκες στα ψηφοδέλτια. Όσο περισσότερο, όσο περνάνε τα χρόνια που είμαι δηλαδή στην επιχείρηση και στην πολιτική, εγώ είμαι όλο και περισσότερο υπέρ των ποσοστώσεων. Διότι έχω την εντύπωση ότι αν πούμε, τώρα, κοιτάξτε αυτό είναι άκαμπτος μηχανισμός και υπάρχουν γυναίκε οι οποίε δεν διαθέτουν απαραίτητα προσόντα κλπ. Όλα αυτά είναι σαν χλαμάρες. Ε, χρειάζεται να καλύψουμε τόσα πολλά χρόνια και δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Υπάρχουν διάφορες απεικονίσεις, δηλαδή αν ακολουθήσουμε το φυσικό ρυθμό θα χρειαστούμε άλλα 70 χρόνια για να φτάσουμε εκεί που είναι οι άντρες σήμερα ή 100 χρόνια κλπ. Πάλι ξαναλέω ότι πρόκειται για τεράστια απώλεια. Δεν μπορούμε να την αντέξουμε τέτοια απώλεια ικανοτήτων δηλαδή και όλο και περισσότεροι άνδρες το κατανοούν αυτό σιγά σιγά και στην πολιτική γιατί η Ανιέσκα ζήτησε ας πούμε κάποιες συμβουλές πώς μπορούμε να επιταχύνουμε την διαδικασία ώστε να αποκτήσουν περισσότερες ε, δυνατότητες, ικανότητες, προνόμια οι γυναίκες στην ε, ε, εξουσίες μάλλον στην πολιτική. Και στις επιχειρήσεις υπάρχουν πολλές οργανώσεις, άντρε δηλαδή, που αποφάσισαν ότι για τις επιχειρήσεις τους, για την κοινωνία, είναι καλό να έχουν περισσότερες γυναίκες στα υψηλά επίπεδα της ιεραρχίας. Το ίδιο ισχύει και την πολιτική. Μετά από το κίνημα MeToo ανοίγεται η ευκαιρία για μας να χρησιμοποιήσουμε τον αγώνα αυτό διότι ο κόσμος γενικά μας υποστηρίζει περισσότερο τώρα την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών. Ο κόσμο θέλει όντω περισσότερε γυναίκε στην πολιτική, περισσότερε γυναίκε στι επιχειρήσει ε, και αισθάνονται πλέον άνετα με την προοπτική αυτή. Άρα να προχωρήσουμε. Μην είστε ντροπαλέ, να κάνουμε τη δουλειά μα, να ολοκληρώσουμε τι συζητήσει μα, διότι πρέπει να το κάνουμε για τι οικογένειέ μα, για τι κοινωνίε μα, για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι όσο περνούμε τον καιρό συζητώ διάφορε ιδέε, χωρίς να προωθούμε τα θέματα αυτά, τόσο περισσότερο θα καθυστερούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θεωρώ ότι η δικτύωση είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας και είναι και ένας τρόπος επίλυσης του προβλήματος. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στη δόκτωρα Μέριλ Κένι, λέκτορα στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας που με προσκάλεσε για να μιλήσω για την ε, Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας. Ε, είμαι ακαδημαϊκός. Ε, θα σας εξηγήσω τι έρευνα έχουμε κάνει για τα εμπόδια που ε, αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, ε, για τη σημασία των ποσοστώσεων και τι έχουμε διδαχθεί από την ε, δική μας κοπιά, τη Σκοτία και το Ηνωμένο Βασίλειο και νομίζω ότι υπάρχουν παραλληλισμοί ε, και με τη δική σας οποιαδήποτε πραγματικότητα. Στην Σκοτία έχουμε γυναίκες στην πολιτική τα τελευταία χρόνια. Η Νίκολα Στέρτζον έγινε η πρώτη Πρωθυπουργό της Σκοτίας το 2014 και διόρισε διάφορες γυναίκες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τα, ε, τα τρία ε, μεγαλύτερα κόμματα ηγούνται από γυναίκες. Έχουμε και πολλές ε, και έχουμε και είχαμε γυναίκες υπουργού από όλα τα κόμματα. Ε, αυτό όμως το νέο πρόσωπο τη σκοτσέζικη πολιτική θα πρέπει να το βάλουμε σε ένα σωστό πλαίσιο. Ότι και στο Ηνωμένο Βασίλειο γενικότερα και πέραν ε, υποεκπροσωπούνται οι γυναίκε. Ο ρόλο ε, ε, τη εκπροσώπηση των γυναικών στο Κοινοβούλιο ε, έχει φτάσει σε ένα πλατό. Ε, 45 γυναίκε έχουμε στο Κοινοβούλιο. Ε, είμαστε στο ίδιο επίπεδο με, τις προηγούμενες, με το προηγούμενο Κοινοβούλιο. Ε, δεν έχουμε ποτέ έγχρωμη γυναίκα στο Σκοτσέζικο Κοινοβούλιο. Ε, Επομένω και στη Σκωτία, ε, και όπως και σε πολλές χώρες, η εικόνα αυτή ε, υπόσχεται πολλά, αλλά δεν, είναι, ε, δεν τα έχουμε καταφέρει 100%. Δεν πρέπει λοιπόν να χάσουμε την ορμή που έχει δημιουργηθεί. Βάζω λοιπόν το ευρύτερο πλαίσιο για την εκπροσώπηση των γυναικών, για την οποία μιλήσατε, και ξέρουμε ότι η υποεκπροσώπηση των γυναικών είναι ένα κλασικό στοιχείο ε, και στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο. Κάτω από 24% των ε, γυναικών είναι στα κοινοβούλια παγκόσμια. Ε, και δεν μόνο η υποεκπροσώπηση, είναι και η υπερεκπροσώπηση των ανδρών στα κοινοβούλια. Πάνω από 75% στα κοινοβούλια είναι άντρες. Και μόνο τρία κοινοβούλια στον κόσμο τα πάνε καλύτερα. Το 2003 η Σκοτία ήταν, αν είχε μπει στην παγκόσμια κατάσταση, θα ήμασταν τέταρτη. Τώρα είμαστε 32η. Έχουμε πέσει δηλαδή. Και το ίδιο συμβαίνει και σε πολλές άλλες χώρες που τα πάνε χειρότερα. Ορισμένες χώρες ε, έχουν επιβάλει διανόμου ποσοστώσεις για να επιταχύνουν πάρα πολύ την εκπροσώπηση των γυναικών. Τι εξηγεί αυτά τα pattern και τι χρειαζόμαστε ούτω ώστε να έχουμε περισσότερες γυναίκες ε, στην πολιτική. Η Πέπε Νόρι και η Κρουκ, ε, που είναι ακαδημαϊκοί και που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, λένε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ε, πολύ καλό συνταγματικό πλαίσιο, αστικά δικαιώματα των γυναικών και ποσοστώσεις στο Σύνταγμα, οι οποίες δίνουν τεράστιες ευκαιρίες για την κινητοποίηση των γυναικών για τα θέματα αυτή της εκπροσώπησης. Ε, σημασία έχουν και τα εκλογικά συστήματα ε, και το πώς επιλέγουν ε, τα κόμματα τι γυναίκες. Βλέπουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των γυναικών, ή μάλλον εκεί όπου έχουμε πολλές γυναίκες, έχουμε και ποσοστώσεις από τα κόμματα και έχουμε δια νόμου υποχρεωτικά νούμερα για την εκπροσώπηση των ε, γυναικών. Αλλά αυτό δεν αρκεί από μόνο του για να αυξήσει την αύξηση της παρουσίας των γυναικών στην πολιτική. Ε, το βασικό εμπόδιο στην ε, πολιτική στις γυναίκες είναι τα πολιτικά κόμματα όμως. Οι γυναίκες μπορεί να αποφασίσουν ότι θέλουν να ε, κατέβουν σε εκλογές, αλλά πρέπει να, επιλεγούν πρώτα από τα πολιτικά κόμματα. Ε, και νομίζω ότι τα πολιτικά κόμματα και όχι οι ψηφοφόροι είναι αυτοί που αποτελούν τους πραγματικούς φύλακες των ε, πολιτικών αξιωμάτων. Δόθηκε μεγάλη προσοχή τα τελευταία χρόνια στι πρωτοβουλίε για να ενθαρρύνουν τι γυναίκε να κατέβουν στην πολιτική μέτρα, όπω κατάρτιση, ε, οικονομική στήριξη, mentoring και σχετικά προγράμματα. Αυτά τα προγράμματα είναι πολύ σημαντικά για να αναπτύξουν το δυναμικό του οι γυναίκε. Αλλά υπάρχει ο κίνδυνο μερικέ φορέ να πούμε ότι το πρόβλημα τη υποπροσώπηση των γυναικών ε, έγκυται στις ίδιες τις γυναίκες. Ανταυτού η έρευνα δείχνει ότι το πρόβλημα το έχουν τα κόμματα. Τα κόμματα δεν επιλέγουν γυναίκες υποψηφίους και δεν επιλέγουν για θέσεις που μπορούν να κερδίσουν. Όταν απαιτείται να επιλέξουν γυναίκες, όπως μέσω ποσοστώσεων, μπορούν να βρουν γυναίκες. Ε, οι ανισότητες στη ζήτηση οδηγούν σε ανισότητες στην προσφορά. Θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγέ στα κόμματα. Είναι σημαντικό να υπάρχουν ποσοστώσει καλοσχεδιασμένε, με το κατάλληλο εκλογικό σύστημα, να εφαρμόζονται σωστά. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Το τελευταίο στοιχείο που θα ήθελα να σα τονίσω πριν κλείσω είναι η θεσμική και κοινοβουλευτική μεταρρύθμιση. Θα πρέπει να διευκολύνουμε ε, τους τρόπους που λειτουργούν τα όργανα αυτά. Ε, να έχουμε μέτρα για την φύλαξη των παιδιών, ε, το πόσες ώρες ε, συνεδριάζει η Βουλή κτλ. Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για να κατέβουν οι Έλληνες στην πολιτική, αλλά για να ξανακατέβουν στην πολιτική. Το σκοτσέζικο κοινοβούλιο έχει αναγνωρίσει ότι θα πρέπει οι ώρες ε, της συνεδρίασης να είναι φιλικές για την οικογένεια, να υπάρχουν να υπάρχει η δυνατότητα για παιδικούς σταθμούς, ε, ούτως ώστε οι μητέρες να δίνουν τα παιδιά τους μέσα κοντά στη Βουλή και να υπάρχουν γενικά φιλικές πρακτικές για την οικογένεια. Αυτό, ε, αυτές, εμείς κάναμε προσπάθειες στη Σκωτία όπου και έρχεται σε αντιπαράθεση με τις πρακτικές στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ε, κανείς για να μπει στο κοινοβούλιο ξεχνάει όλα τα άλλα. Και δεν υπήρχε δυνατότητα ε, μέχρι το 2010 για παιδικό σταθμό για τις γυναίκες ε, πολιτικούς. Θέλουμε να δούμε και να αποδείξουμε, ή μάλλον η αλλαγή μπορεί να γίνει, αλλά χρειάζονται ευκαιρίες. Θα πρέπει να προωθήσουμε με επιχειρήματα την εκπροσώπηση των γυναικών. Η πρόοδος δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη λόγω της ε, σημερινής παρουσίας των γυναικών ε, στην ε, πολιτική. Ε, είπαμε ότι από τότε μέχρι τότε έχουμε τέτοια πρόοδο, αλλά θεωρούμε ότι η πρόοδος είναι γραμμική. Είναι λάθος αυτό. Επίσης, ξέρουμε ότι και στη Σκοτία και αλλού η παρουσία των γυναικών έχει αλλάξει την ποιότητα της νομοθεσίας ε, και το πώς λειτουργεί η πολιτική. Αλλά τα νούμερα δεν τα λένε όλα. Η σχέση είναι περίπλοκη, διαμορφώνεται από το, τις θεσμικές σχέσεις, από τις κομματικές σχέσεις. Τα πολιτικά κόμματα ε, γενικά δείχνουν μεγαλύτερο και άνοιγμα στις ανησυχίες ε, των γυναικών, αλλά δεν αρκεί αυτό. Οι ποσοστώσεις είναι η πιο αποτελεσματική στρατηγική για να αυξηθεί η εκπροσώπηση των ε, γυναικών, αλλά δεν αρκεί να το κάνουμε μια φορά. Θα πρέπει να υπάρχει συνεχής δέσμευση και δράση από τα πολιτικά κόμματα. Θα πρέπει να καλοσχεδιάζουν τις ε, κυρώσει και να υπάρχουν τις ποσοστώσεις και να υπάρχουν και κυρώσει για όσου δεν τι εφαρμόσουν. Και μπορεί να υπάρξουν βεβαίω και προβλήματα σε αυτή την πορεία. Χρειάζονται οι ποσοστώσεις και χρειάζονται και πολλές άλλες ε, μεταρρυθμίσεις. Χρειάζεται λοιπόν μια συνολική στρατηγική. Ευχαριστώ την κυρία Κέλλη. Οι ποσοστώσεις μαζί με την πολιτική βούληση μπορεί να βοηθήσει. Τώρα επιτρέψτε μου να αρχίσουμε τη συζήτηση, να ε, αρχίσω τη συζήτηση, δίνοντας το λόγο στα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Θα προσπαθήσω να δώσω το λόγο σε όσο το δυνατόν περισσότερες εθνικές αντιπροσωπείες. Όμως σημειώστε ότι έχουμε μόνο 35 λεπτά στη διάθεσή μας. Θα παρακαλέσω λοιπόν όλες και όλους τους συμμιλητές να περιοριστούν σε δύο λεπτά. Πρώτος ομιλητής ή πρώτη ομιλήτρια, η κυρία Μάρτα Ματράικ από την Ουγγαρία. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμού των γυναικών βουλευτών από το Εθνικό μας Κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό να δώσουμε μια καθαρή εικόνα της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική και στην κοινωνία. Στην Ουγγαρία θεωρούμε ότι πολιτικά, κοινωνικά, ανθρώπινα και απόψη δικαίου δεν υπάρχει πολύ καμία διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλλα. Αυτή την αρχή την περιλαμβάνει στο άρθρο 15 παραγραφος 3 και το Ουγγρικό Σύνταγμα. Λέει ότι είναι απόλυτα ίσα τα δύο φύλλα. Βέβαια, η φύση προβλέπει διαφορετικές, ε, με σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι γυναίκες ανέκαθεν έχουν <clears throat> αναμειχθεί στην τοπική πολιτική. Εμείς δεν πιστεύουμε τόσο πολύ στις ποσοστώσεις. Θεωρούμε ότι σημαντική είναι η στήριξη των ταλέντων των γυναικών για να παίξουν ρόλο και στην κοινωνία και στην πολιτική. Στην Ουγγαρία όλο και περισσότερες γυναίκες καταλαμβάνουν μεσαίες και υψηλότερες ε, θέσεις ευθύνης. Στην τοπική αυτοδιοίκηση ε, αριθμούμε πολλές γυναίκες δημάρχους, αναπληρωτές, ε, αναπληρώτριες μάλλον δημάρχους και σε άλλες θέσεις. Σήμερα το δημογραφικό πρόβλημα είναι κοινό σε όλη την Ευρώπη. Ορισμένοι βλέπουν την λύση στο μεταναστευτικό και, το, και υποστηρίζουν τη μεταναστευσή. Η, Ουγγρική, η Ουγγαρία μάλλον βρίσκει ε, τη λύση αυτή ότι δεν είναι η κατάλληλη. Δίνουμε περισσότερο στήριξη στι ουγγρικέ οικογένειε, ώστε να γεννηθούν περισσότερα παιδιά, να μπορέσουν να βρουν δουλειά και οι γυναίκε να μπορούν και να βρουν δουλειά, αλλά και να ε, αναμειχθούν στην πολιτική. Για μένα, η γυναίκα έχει μια ιδιαίτερη προσωπικότητα και ιδιαίτερη ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, που πρέπει να μπορέσει με τον τρόπο αυτό να εμπλουτίσει και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Ματράη. Η κυρία Ζωρόφσκα από την Πολωνία. Έχετε το λόγο, κυρία μου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σας απευθύνω πρώτα-πρώτα ε, την καλημέρα μου και θα ήθελα να αρχίσω με ένα αισιόδοξο μήνυμα. Εκπροσωπώ την Πολωνική Γερουσία και προέρχομαι από μια περιοχή όπου 75% των γυναικών, δηλαδή μάλλον 75% των γυναικών στην Πολωνική Γερουσία, ε, είναι μέλη δηλαδή, στην Πολωνική Γερουσία. Ε, πρώτη γυναίκα που προείδρευσε την τοπική βουλή της Σιλεσίας. Τότε την είχαν χαρακτηρίσει αυθάδη την πρώτη αυτή ε, πρόεδρο. Αλλά μπόρεσε να επιτύχει πολλά πράγματα. Οργάνωσε τις γυναίκες, έγραφε άρθρα και εγχειρίδια και γενικώ προκαλούσε αναστάτωση. Αυτά έλεγαν για αυτήν. Όταν δεν προκαλούσε αναστάτωση, ωστόσο, συνέβαλε στην ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στην Πολωνία. Έχουμε κοντά μα ένα θαυμάσιο παράδειγμα, την κυρία Χενρίκα Μπόχνιαρτ, από τι πρώτε γυναίκε, μίλησε προηγουμένω. Πολωνέ που οργάνωσε την δράση, όπως αυτή που σας εξήγησε, του Πολωνικού Κογκρέσου των Γυναικών. Βέβαια, μην νομίζετε ότι η εικόνα είναι τόσο ρόδινη. Υπάρχουν αριθμοί που δείχνουν ότι η εκπροσώπηση των γυναικών στο Κοινοβουλίο, στην Κάτω Βουλή, αλλά και στην Άνω Βουλή, αλλά και στις τοπικές κυβερνήσεις, στις ε, τοπικές αυτοδιοίκησεις δηλαδή, δείχνουν τα νούμερα αυτά ότι χρειάζομαστε 60 χρόνια ακόμα για να έχουμε ισότιμη εκπροσώπηση με τους άντρε. κυρία από την Πορτογαλία. Καλημέρα σε όλου. Ε, θα μιλήσω στα πορτογαλικά που είναι η μητρική μου γλώσσα, οπότε θα ήθελα να σα βάλω να βάλετε τα ακουστικά σα. Θα, για να ενισχύσουμε την εκπροσώπηση των γυναικών τότε θα πρέπει να αυξήσουμε τον αριθμό των γυναικών. Δηλαδή το 2017 ε, ε, είχαμε ποσοστά με, κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες οι οποίες ε, άρχισαν να αυξάνονται, έφτασαν το 1980 δηλαδή το 6,4 μετά το 6,2 και ε, το 2006 φτάσαμε στην θέσπιση μιας νομοθεσίας η οποία ε, προέβλεπε ελάχιστη εκπροσώπηση 33% ε, των γυναικών στους εκλογικούς καταλόγους των διαφορετικών πολιτικών κομμάτων και για τις εθνικές εκλογές και για τις ευρωεκλογές. Μετά λοιπόν από αυτή την έγκριση καταφέραμε να έχουμε πράγματι ένα τρίτο των θέσεων στο Εθνικό Κοινοβούλιο ως γυναίκες. Άρα λοιπόν ακόμα και έτσι τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ χαμηλά, δηλαδή τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλά ο, και έτσι το, η δική μας κυβέρνηση πρότεινε να υπάρξει ελάχιστη εκπροσώπηση των γυναικών στον κοινοβούλιο του τάξης του 40% ε, και θεωρούμε πως ε, αφού θα έχει περάσει ήδη γιατί το νομοσχέδιο κατατέθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο ε, θα ισχύσει και για τις επόμενες ευρωεκλογές. Εδώ βλέπουμε λοιπόν μια πολύ σημαντική διάσταση ε, σε ό,τι αφορά αυτή την επίτευξη του 40% και αυτό τι είναι δηλαδή επιβολή κυρώσεων ε, προκειμένου ε, πράγματι να επιβληθεί αυτό το ελάχιστο 40%. Όμως για να επιτύχουμε την ισόρροπη εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική εξουσία θα πρέπει να κάνουμε και περισσότερα. Δηλαδή εκείνο που θα πρέπει να δούμε είναι ε, ολοένα και περισσότερες ε, γυναίκες οι οποίες ε, περιλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους, στους υποψηφίους. Γιατί στην πραγματικότητα σήμερα αυτό που συμβαίνει είναι ότι ακόμα και αυτές οι γυναίκες που εκλέγονται και επιλέγονται, επιλέγονται από άνδρες. Άρα λοιπόν δεν θεωρούμε ότι θα, με μια απλή αλλαγή της νομοθεσίας θα επιτύχουμε όλα εκείνα που θέλουμε. Δηλαδή θα πρέπει να δώσουμε περισσότερες δυνατότητες για τις γυναίκες προκειμένου να μπορούν να εκλέγονται. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, thank ε, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ταβάρες. Ε, η κυρία ε, Μαρή Πενερικουσόν από τη Γαλλία έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που εκπροσωπώ την ε, Γαλλία σήμερα εδώ με την ευκαιρία της Διεθνούς ημέρας της γυναίκας που οργανώνεται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική ζωή από τις πιο μικρές κοινότητες μέχρι τα υψηλά επίπεδα για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική. Διότι είμαι και πρόεδρος της αντιπροσωπείας των γυναικών στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Η ισότητα των φύλων περιλαμβάνεται από αιώνες στο Σύνταγμά μας. Με διαρκή νομοθέτηση εξασφαλίζεται και η επιχειρησιακή ισότητα τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί πολύ ισχυρά οι γυναίκες και στην πολιτική συζήτηση. Η κυβέρνησή μας μαζί με το κοινοβουλίο μας ασκούν την πολιτική αυτή, για παράδειγμα μέσω και του νέου προσώπου της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης που έχει πολύ ισχυρό το γυναικείο στοιχείο με 48% των γυναικών βουλευτών. Δηλαδή βουλευτών είναι στη, στην δική μου δηλαδή κοινοβουλευτική ομάδα που είναι η Δημοκρατία ε, εν πορεία, ε, Ρεπιμπλίκα Μάρς. Ενισχύουμε τους στόχους της ισότητας και διαπιστώνουμε βεβαίως ότι σε άλλους τομείς οι γυναίκες αριθμητικά υστερούν. Χρειάζεται σημαντική ε, προώθηση των ε, ε, δικαιωμάτων των γυναικών. Χρειάζεται να καλυφθούν δεκαετίες και αιώνες καθυστερήσεων. Θα πρέπει να είμαστε απολύτως αδιάλακτες σε αυτό και θα καταλήξω με ένα παράθεμα του Λαμπτεγκούς. Η... Δεν, το, το Σύνταγμα δεν μπορεί να είναι ισχυρό εάν η πλειοψηφία των πολιτών, που είναι γυναίκες δηλαδή, δεν έχουν συμμετάσχει στη σύνταξή του. Ευχαριστώ. Τώρα η κυρία Βικτόρια Σμιλίτα Λίνσα από την Λιθουανία. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, εκπροσωπώ το Λιθουανικό Κοινοβούλιο, όπου είμαστε οι γυναίκες λιγότερο από 25% των μελών. Και ομολογώ ότι ζηλεύω κάπως το, την ε, Ισπανίδα συναδελφό μου που είπε προηγουμένως ότι έχουν 67% γυναίκες υπουργού στην κυβέρνηση. Εμείς έχουμε 0%. Ελπίζω ότι είναι προσωρινό αυτό. φοβούμε όμως ότι στην πραγματικότητα είναι, ε, μπαίνει σε, σε μια μεγαλύτερη εικόνα. Ένα από τα προβλήματα που βλέπουμε συχνά είναι ότι οι γυναίκες που εκλέγονται στα κοινοβούλια, νεαρές πολιτικοί δηλαδή, τείνουν να ασχολούνται με ελαφρότερα γυναικεία θέματα και έχουν δυσκολία έτσι να φτάσουν στα ηγετικά ε, επίπεδα. Όσο ανεβαίνεται δηλαδή την ιεραρχική κλίμακα, όλο λιγότερο οι γυναίκες βρίσκεται. Κάτι άλλο που έχουμε δει τελευταία είναι ότι με το κίνημα Me Too, ακόμα και οι γυναίκες δημοσιογράφοι που έγραψαν για το θέμα αυτό, αντιμετώπισαν απειλές. Και πολύ άσχημες συμπεριφορές. Cyberbullying δηλαδή, bullying μέσω του διαδικτύου. Μόνο και μόνο επειδή έγραψαν για τα πράγματα αυτά και έδειξαν ενδιαφέρον. Και αυτό και αυτέ οι απειλέ δεν προέρχονται μόνο από άνδρε, αλλά φαίνεται πω προέρχονται και από γυναίκε. Διερωτώ λοιπόν, τι λάθος κάνουμε. Νομίζω ότι ενώ η Ευρώπη είναι θαυμάσια ήπειρος για να είναι κανείς η γυναίκα, μένουν ακόμα, ακόμα πολλά πράγματα να γίνουν. Και θα ζητήσω και από τους άνδρες να συμμετάσχουν πολύ εντονότερα για την επίλυση του θέματος, διότι δεν, κάτι τέτοιο δεν θα ενισχύσει μόνο τη θέση των γυναικών, θα ενισχύσει συνολικά την κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα η κυρία Μαριέλα Αριστίδου από την Κύπρο σας, στην Κύπρο γίνονται μικρά και σταθερά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Εν τούτης, παρά την αυξανόμενη ενεργό συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική και δημόσια ζωή, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε σημαντικές θέσεις λήψης αποφάσεων στην κυβέρνηση, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια. Θα ήθελα να επισημάνω ωστόσο ω θετική εξέλιξη το διορισμό γυναικών από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε σωρία υψηλόβαθμων θέσεων. Επί του παρόντο, οι Κύπριε γυναίκε αναλαμβάνουν δυσανάλογο μερίδιο του νοικοκυριού, τη φροντίδα των παιδιών και των οικογενειακών ευθυνών. Συναφώ, είναι επίγουσα ανάγκη να εντατοικοποιηθούν οι προσπάθειε για την καλύτερη συμφιλίωση τη επαγγελματική και οικογενειακή ζωή μέσω τη παροχή προσιτών και ποιοτικών υπηρεσιών, οι οποίε θα είναι φιλικέ προ την οικογένεια και την παιδική μέρημνα. Θα ήθελα όμω να κάνω και ιδιαίτερη μνήα στα θετικά μέτρα που έλαβε πρόσφατα η Κυπριακή κυβέρνηση ω προ την εσωμάτωση τη διάσταση του φύλου σε όλε τι πολιτικέ. Το Υπουργικό Συμβούλιο υιοθέτησε οδηγό ένταξη τη διάσταση του φύλου στι δημόσιε πολιτικέ με στόχο την ευαισθητοποίηση των στελεχών τη δημόσια διοίκηση που λαμβάνουν μέρο στη διαδικασία χάραξη πολιτική, στην κατάρτιση των προπολογισμών και στο προγραμματισμό δράσεων που αφορούν στη διάσταση του φύλου. Επίση, πρόσφατα συντάχθηκε οδηγό υπέρβαση του γλωσσικού σεξισμού στη γλώσσα των εγγράφων τη δημόσια διοίκηση τη Κυπριακή Δημοκρατία. Χαιρετίζω τέλο την πρόσφατη απόφαση της Κυπριακής Κυβέρνησης για ενσωμάτωση σε συστηματική βάση της διάσταση του φύλου σε ολόκληρο το φάσμα ενάσκηση τη εξωτερική πολιτική του κράτους, συμβάλλοντα κατά αυτόν τον τρόπο στι διεθνεί προσπάθειες για εξάλληψη των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλου του τομεί και για εντατικοποίηση τη προόδου προ αυτή την κατεύθυνση. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κριστίνα Γιουρισνίτη από τη Ρουμανία έχει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, αποτελεί η τιμή μου να συμμετέχω στη σημερινή διακοινοβουλευτική συνεδρία στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας ε, ε, του 2019. Ωστόσο, ε, θα ήθελα να μιλήσω στα γαλλικά να συνεχίσω την παρέμβασή μου καθώς είμαι και καθηγήτρια γαλλικών. Ε, για την ισότητα των ευκαιριών ε, στον πολιτιστικό τομέα, θα ήθελα να πω δύο λόγια. Θα ήθελα να μιλήσω να, να μιλήσω για το θέμα της στήριξης των γυναικών για να μπορέσουν να μπουν στην πολιτική. Εκπροσωπώ τη Ρουμανία. Είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας Ευκαιριών της Εθνικής μας Βουλής, του Εθνικού μας Κοινοβουλίου. Εμείς έχουμε εκλογές σε δύο χρόνια. Οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι το 52% του συνολικού πληθυσμού. Η εκπροσώπησή τους όμως ε, στο Κοινοβούλιο είναι πολύ κάτω του ποσοστού αυτού. Βρίσκεται στο 18% μόνο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είμαστε στο 36,2%. Αυτό είναι το ποσοστό των ε, γυναικών πολιτικών. Εμείς είμαστε στο 18%. Ε, μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, φτάσαμε παρόλα αυτά σε αυτό το ποσοστό, που είναι ρεκόρ για μας. Ε, γιατί ε, στην Γερουσία ε, η εκπροσώπηση των γυναικών φτάνει μόνο στο 11%. Εγώ πρότεινα, ο, υπό την οδειότητά μου της Πρόεδρου της Επιτροπής Ισότητας Ευκαιριών και Γυναικών, να προτείνω, πρότεινα λοιπόν υποχρεωτικές ποσοστώσεις μίνιμουμ 30% γυναικών στα ψηφοδέλτια, στις ε, αυτοδιοικητικές εκλογές αλλά και στις ε, βουλευτικές εκλογές. Αυτό έχει προταθεί όχι μία φορά, πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Αλλά δεν υπήρχε η απαραίτητη πολιτική στήριξη για να περάσει. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είπε ότι στην Ευρώπη έχουμε κοινέ αξίες και ισότητα ευκαιριών. Πολύ σύντομα, κατά πάσα πιθανότητα, η κυρία Κουβεσί θα ε, ανήκει στο προσωπικό της Ευρωπαϊκής εισαγγελία. Είναι η πρώτη Ρουμάνα ε, εισαγγελέας. Ε, ξέρουμε από έρευνες ότι όσο περισσότερες γυναίκες έχουμε σε υψηλές θέσεις, ε, τόσο καλύτερη κοινωνία. Είμαι υπέρ των ποσοστώσεων στην ε, ρουμανική πολιτική και ελπίζω να ενσωματωθούν και στον εκλογικό νόμο. Υπάρχει ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκδόθηκε στις 15 Ιουνίου για τις ποσοστώσεις. Ε, καταλαβαίνουμε ποιες, ποια είναι τα ωφέλη των ποσοστώσεων για όλους μας, όχι μόνο για τις γυναίκες και τα κορίτσια. Φυσικά αυτό είναι σημαντικό για όλους γιατί οι γυναίκες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Η ε, κυρία Μαρία Καλαρίτη τώρα από την Ελλάδα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, είναι κοινό τόπο ότι και στην Ελλάδα και στην πλειοψηφία της Ευρώπης ε, η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων όχι απλά δεν είναι ισότιμη αλλά είναι εξαιρετικά χαμηλή. Θα τολμούσα να πω ότι μιλάμε για μια πολιτική περιθωριοποίηση που, ε, η οποία συνυπάρχει με την νομική, είναι αντίφαση αυτό βέβαια με την νομική ε, ε, ισότητα. Πριν αναφερθώ στους τρόπους για την ενίσχυση των γυναικών στην πολιτική, θεωρώ ότι αρκετά σημαντικό είναι να μιλήσουμε για το διαχωρισμό μεταξύ της πολιτικής συμμετοχής και της πολιτικής αντιπροσώπευσης στις δομές εξουσίας. Και αυτό γιατί. Γιατί στην πολιτική αντιπροσώπευση δεν συμμετέχουμε απλώς για να διαμορφώσουμε πολιτική ατζέντα, αλλά διαμορφώνουμε στην πολιτική ατζέντα με βάση, τη διαμορφώνουμε με βάση την ατζέντα φύλου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ενσωματώνουμε τη διάσταση του φύλου στις δημόσιες πολιτικές. Άρα δεν θέλουμε περισσότερο μόνο γυναίκες, αλλά θέλουμε και γυναίκες που μπορούν να θέτουν την ατζέντα φύλου στην πολιτική. Έρχομαι τώρα στους τρόπους ενίσχυσης της εξουσίας των γυναικών, στην πολιτική συμμετοχή δηλαδή. Ε, συμφωνώ ότι τα συστήματα ποσοστώσεων αποτελούν το βασικό αλλά όχι το αποκλειστικό εργαλείο για να συμβάλλουν στην επιτάχυνση της ισότιμης συμμετοχής. Απαιτούνται επιπλέον μέτρα. Για παράδειγμα, θέλουμε πιο στοχευμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες, μέτρα και κίνητρα. Θα μπορούσαμε, αν είχαμε χρόνο, να αναφέρουμε και συγκεκριμένα παραδείγματα. Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί παραλείπουμε ε, το, ε, την επιτάχυνση της προόδου στην εξισορρόπηση εργασιακού, προσωπικού, οικογενειακού βίου, γιατί όλες οι έρευνες μας δείχνουν ότι εκεί έχουμε τα μεγαλύτερα έμφυλα χάσματα, στη χρήση δηλαδή του χρόνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αυξήσουμε τις δομές για τη φροντίδα παιδιών εξαρτημένων μελών κτλ. Συμφωνώ απόλυτα με τις προτάσεις γι' αυτό και στο Κοινοβούλιο, αλλά θα έλεγα και γενικότερα. Στην Ελλάδα καταφέραμε, και τελειώνω συγγνώμη, να αυξήσουμε το ποσοστό από το 1 τρίτο στα 40% και στις αυτοδιοικητικές εκλογές το ψηφίσαμε, θα εφαρμοστεί τώρα και ε, ε, αύριο ψηφίζουμε και την αύξηση από το 1 τρίτο στα 40% και στις βουλευτικές εκλογές. Τέλος, θα συμφωνήσω ότι ο ρόλος των κομμάτων, των πολιτικών κομμάτων είναι κέραιο στην αύξηση της ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών. Το διαπιστώνουμε όταν το βλέπουμε στις λίστες που μειώνεται ο αριθμός αντί να αυξάνεται και θα έλεγα να δούμε μέτρα όπως η χρηματοδότηση, να το συνδυάσουμε με χρηματοδότηση κομμάτων και άλλα μέτρα που θα αναφερθώ σε άλλη έλλειψη χρόνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Uh, ευχαριστώ πολύ την κυρία Τελαρίτη και η κυρία Καρδίνα Μέγερ έχει το λόγο τώρα από τη Δανία και θα ήθελα να παρακαλέσω όλους όσους παίρνουν το λόγο να μιλούν μόνο για δύο λεπτά ούτως ώστε να προλάβουμε να ολοκληρώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να παρευρεθούμε σήμερα εδώ. Ε, σε ό,τι αφορά την ισότητα των φίλων, εμείς ε, ε, θεωρούμε πως έχουμε αναλαμβάνει πραγματικά ηγετικό ρόλο ή τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να μας βλέπουμε, αλλά δεν ισχύει αυτό ε, σήμερα και εδώ αναφέρομαι ε, σε ό,τι αφορά το κοινοβούλιο της Δανίας ότι η γονική άδεια, η είναι σήμανο για το 10% ενώ στη Σουηδία, στην ε, Νορβηγία ε, και σε άλλες χώρες ε, γειτονικέ μα είναι ψηλότερα αυτά τα ποσοστά. Ενώ μόνο το 19% είναι γυναίκε στα διευθυντικά συμβούλια. Και συνεχίζουμε να έχουμε και υψηλό μισθολογικό χάσμα στην Δανία και μόνο το 1 τρίτο ε, των ε, βουλευτών είναι γυναίκε στο Εθνικό μα Κοινοβούλιο. Εξακολουθούν λοιπόν να υπάρχουν τέτοιου είδου προβλήματα, αλλά η κυβέρνησή μα είναι πολύ ε, δύσπιστη και δεν επιθυμεί να επιβάλλει ποσοστώσει. Και βασίζεται εδώ σε ένα επιχείρημα ότι θα πρέπει να υπάρχει ελευθερία της επιλογής. Δηλαδή θα πρέπει να μπορεί κανείς να επιλέγει ασχέτως οποιοδήποτε άλλου παράγοντα. Δηλαδή αυτή η έννοια της ελευθερίας βασίζεται στο ακριβώς να μπορεί να επιλέγει κανείς ό,τι επιθυμεί. Αλλά νομίζω πως ε, θα πρέπει να επανεξετάσουμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε αυτή την έννοια ε, της ελευθερίας. Ε, γιατί πραγματικά δεν είναι πραγματικά ελεύθερη μια γυναίκα όταν αντιμετωπίζει τέτοιου είδους δομικούς περιορισμούς και στις δυνατότητες της. Δηλαδή όταν δεν έχει τη δυνατότητα να εκλεγεί δεν νομίζω πω ισχύει δηλαδή αυτή η ελευθερία όταν για παράδειγμα η πρώτη πρωθυπουργό που εξελέγει στη Δανία έλαβε ερωτήσει του τύπου ε, πώς καταφέρνετε να φροντίζετε και τα παιδιά στο σπίτι. Θα πρέπει λοιπόν να επανεξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την έννοια τη ελευθερία και με βάση αυτή την αναθεώρηση να προβούμε στη θέσπιση νομοθεσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ε, την κυρία Μέγερ. Τώρα η κυρία Ελίζα Γκρόσμαν από την Αυστρία έχει το λόγο. Ε, εγώ από την πλευρά μου εκπροσωπώ το Αυστριακό Κοινοβούλιο, ε, το οποίο σε σύγκριση ε, με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σχετικά υψηλή εκπροσώπηση των γυναικών και υπάρχουν βέβαια και δεσμευτικέ ποσοστώσει οι οποίε ισχύουν στου εκλογικού καταλόγου διαφόρων ε, πολιτικών κομμάτων, αλλά α μην ξεχνάμε ότι για να περιληφθεί κανεί στον εκλογικό κατάλογο ενό πολιτικού κόμματο, ε, όχι μόνο προεπιλέγεται, αλλά θα πρέπει να έχει και ένα ε, ιστορικό πολιτικό, συμμετέχοντα δηλαδή σε οργανισμού τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, σε, σε δήμου και κοινότητε και ούτω Άρα αυτό τι σημαίνει, ότι τα μέτρα που λαμβάνουμε θα πρέπει να επεκταθούν και σε όλους εκείνους τους ε, τομείς. Στις διάφορες δηλαδή πολιτικές βαθμίδες. Γιατί και εγώ για παράδειγμα μέσω του Δημοτικού μου Συμβουλίου και της εκλογής μου εκεί κατάφερα να περάσω ε, στον ε, πολιτικό κόσμο και στα Δημοτικά Συμβούλια η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τις γυναίκες γιατί η κατανομή αν θέλετε των ρόλων εκεί είναι πολύ πιο παραδοσιακή από ό,τι αλλού. Άρα λοιπόν οι λίγε γυναίκε οι οποίε ε, συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο συχνά είναι αρμόδιε για παράδειγμα ε, για να, γίνουν τα, να ψήσουμε τα μπισκότα ή να οργανώσουμε τι διάφορε εκδηλώσει. Ε, και αυτό βέβαια αποθαρρύνει πολλέ γυναίκε από το να θέλουν να συμμετάσχουν στην πολιτική όταν βλέπουν να τους κατανέμεται ένας τόσο υποτιμητικός παραδοσιακός ρόλος. Ε, εμείς λοιπόν ως γυναίκες σοσιαλδημοκράτες ε, επιθυμούμε να ληφθούν τα κατάλληλα εκπαιδευτικά μέτρα όχι επειδή η εκπαίδευση που λαμβάνουν οι γυναίκε, αλλά αντιθέτω προκειμένου να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθηση των γυναικών, έτσι ώστε οι γυναίκε λοιπόν να τολμούν, να κάνουν περισσότερα και να αντιμετωπίζουν τσαραλέα τον ανταγωνισμό από τους άνδρες. Σας ευχαριστώ ε, πραγματικά ε, θερμά για τις ε, ε, σημερινές συζητήσεις που κάνουμε και εύχομαι ό,τι καλύτερο για το κοινοβούλιο σας και τα υπόλοιπα κοινοβούλια ε, προκειμένου να επιτύχουμε μια πιο ισότιμη, πιο δίκαια κοινωνία. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γκρόσμαν. Ευχαριστώ. Η βαρόνη Τζένιφερ Άντερσον από το Ηνωμένο Βασίλειο. Μικρόφωνο παρακαλούμε, την ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Φαίνεται ότι είμαι καινούργια εδώ, ε. Ακούσαμε για αυτό το ποσοστό 36% για το Σκοτσέζικο Κοινοβούλιο. 36% γυναίκες. Στη Βουλή των Κοινοτήτων το ποσοστό είναι 32%. Ε, ήμουνα στην ε, Ουαλική ε, Βουλή, η οποία δημιουργήθηκε το 1999. 12% ε, 12 χρόνια. Ξεκίνησε με 50% υποχρεωτική εκπροσώπηση των γυναικών, κάποια στιγμή το ξεπεράσαμε. Ε, ήμουνα ε, αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση και ήμουν και στο Υπουργικό Συμβούλιο και πάνω το 50% ήταν γυναίκες. Τώρα όμως ε, έχει υποχωρήσει η εκπροσώπηση των γυναικών, έχουμε πάει στο 42%. Αυτό που είναι ενδιαφέρον όμω είναι πώς επετεύχθη αυτό το υψηλό ποσοστό των γυναικών και πώς θα συνεχίσουμε το διατηρούμε. Καταρχάς, υπήρχαν ποσοστώσει ε, για τα δύο βασικά κόμματα. Και το τρίτο κόμμα επίσης είχε πολύ θετική δράση υπέρ των γυναικών. Είναι μεικτές οι εκλογικές περιφέρειες, έχουμε συστήματα με εκλογικούς καταλόγους και υπάρχει λοιπόν μια μορφή ε, αναλογικότητα στην εκπροσώπηση και αυτό βοήθησε. Όμως, ε, αυτό που έχει σημασία είναι ότι χάρη στην ε, συμμετοχή μας ε, άλλαξε ο τόνος, άλλαξαν τα θέματα συζήτησης. Η απογοήτευση ήταν τα ΜΜΕ. Από την αρχή παρατηρήσαμε ότι το BBC ήθελε να καλύπτει μόνο ε, τους διχασμούς, ε, τους καυγάδες και τις διχόνοιες, ε, επικεφαλής των οποίων πάντα ήταν σχεδόν οι άντρες. Ευχαριστώ την κυρία Άντερσον. Η κυρία Αλεσάνδρα Μαϊολίνο από την Ιταλία. Κυρία Μαγιορίνο. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ενημερώσω όλους για την σημερινή κατάσταση σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων στην Ιταλία. Το σημερινό κοινοβούλιο είναι ένα κοινοβούλιο όπου έχουμε τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση που είχαμε ποτέ ε, των γυναικών. Έχουμε φτάσει στο 34%. Δεν είναι καταπληκτικό, αλλά είναι βελτίωση. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ιταλικής Δημοκρατίας υπάρχει πρόεδρος της Γερουσίας της Ιταλίας. Υπάρχουν και πιο αυστηροί νόμοι για την καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών και της γυναικοκτονίας. Όμως, οι εποχές που ζούμε είναι δύσκολες. Στην Ιταλία και ίσως και παντού. Τα δικαιώματα των γυναικών που θεωρούσαμε ότι ήταν κεκτημένα, αμφισβητούνται. Το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, ε, σε ό,τι αφορά την εγκυμοσύνη, στην πρόσβαση στην ε, αντισύλληψη. Αφισβητείτε. Ακούγονται πάρα πολλοί να λένε ότι η φυσική θέση της γυναίκας είναι το σπίτι. Και ότι μόνο όταν γίνει μητέρα αισθάνεται ότι ολοκληρώνεται. Ότι γεννιέται για να γίνει μητέρα. Αυτό είναι το πεπρωμένο της αυτές οι δηλώσεις θεωρούσαμε ότι ήταν του παρελθόντος, ότι είναι ξεπερασμένες. Κάνω έκκληση λοιπόν σε όλους σας να σταθείτε ενωμένοι, γιατί μας περιμένουν πάρα πολλά ακόμα, πολλές μάχες, πολλές προσπάθειες και σας καλώ να στηρίξετε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πολεμήσει αυτές τις ε, δυνάμεις που θέλουν να μας πάνε πίσω στο παρελθόν για να πετύχουμε την ισότητα και για να αναπτύξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις κοινωνίες μας. Ευχαριστώ. Τρεις ομιλήτριες μας μένουν. left, but... Αλλά βέβαια δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα παρακαλέσω λοιπόν τις τρεις ε, να απομένουν ομιλήτρες να μιλήσουν μόνο για ένα λεπτό η καθεμία. Πρώτη, η κυρία Εύα Ματίας από την Τσεχία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου μια πολύ σύντομη λοιπόν τοποθέτηση εκ μέρους μου. Οι οργανώσεις που ασχολούνται με την πολιτική των φίλων σε όλα τα επίπεδα ε, έχουν μεγάλη σημασία. Η σημερινή μας συνάντηση είναι σημαντική επίσης, κυρίως διότι επιτρέπει ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ γυναικών, έτσι ώστε να ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους. Διότι οι γυναίκες με αυτοπεποίθηση είναι αυτές που χρειάζονται για να μπορέσουν να ομιλήσουν σε συναθρήσεις όπου συνέρχονται πολλοί άνδρες. Διότι οι άνδρες εκείνοι πρέπει να κατανοήσουν πρώτα-πρώτα ότι χρειαζόμαστε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών. Και ότι ήδη έχουμε φτάσει στο στάδιο αυτό που απαιτείται δηλαδή αυτό. Αυτό πρέπει να φανεί και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια και στην πολιτική. Και νομίζω ότι σε ορισμένες χώρες αυτή η ισότιμη μεταχείριση έχει επιτευχθεί, σε άλλες όχι. Ευχαριστώ πολύ και για την τήρηση του χρόνου. Η κυρία Γερμάνα Ροκά από την Πορτογαλία. Καλημέρα σε όλου. Η ανάγκη του να αλλάξουμε τι νοοτροπίε, ούτω ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν και νέε θέσει οι γυναίκε στη δημόσια ζωή, χρειάζεται και μια αλλαγή τη νοοτροπία. Χρειάζεται δηλαδή περισσότερη ευαισθητοποίηση για το ρόλο των ε, γυναικών σε, σε θέσει ε, κλειδιά προκειμένου δηλαδή στην πραγματικότητα ε, ε, η ε, ανάληψη τέτοιων θέσεων. Αυτό με τη σειρά του απαιτεί προϋποθέτει συγκεκριμένες στρατηγικές οι οποίες θα προωθούν αυτή την πιο ισότιμη προσώπηση των γυναικών. Η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή στην Πορτογαλία έχει αρχίσει να αυξάνεται από το 1974, συγκεκριμένα τις 25 Απριλίου. Ε, δηλαδή, ε, από εκεί και μετά η θέσπιση σχετική νομοθεσία ε, για ελάχιστε ποσοστώσει για την ισότητα των φύλων αποτέλεσε ένα ε, ε περαιτέρω βήμα. Παρότι λοιπόν στην νομοθεσία σήμερα προβλέπουμε την ισότητα και τι ίσε ευκαιρίε ανάμεσα στα δύο φύλλα, η εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική ζωή δεν είναι η, η ενδεδειγμένη. Δεν αντιπροσωπεύει δηλαδή την εκπροσώπηση των γυναικών στην κοινωνία. Ε, και θα πραγματικά αυτό οφείλεται σε νοοτροπίε οι οποίε ακόμα δεν έχουν αλλάξει. Γιατί μόνο με αυτή την αλλαγή θα μπορέσουμε να επιτύχουμε την ε, κατάλληλη εκπροσώπηση των γυναικών. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε πολύ. Τελευταία η κυρία Πέρκοβιτ από την Κροατία. Ορίστε κυρία μου. Θα μιλήσω καλύτερα στο επόμενο πάνελ, διότι είναι πολύ λίγο ο χρόνο. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλες τις βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Μας μένει λίγος χρόνος για τα τελικά σχόλια των προσκεκλημένων μας. Εάν είναι δυνατό, δύο λεπτά για κάθε τοποθέτηση. Αρχίζουμε την κυρία Μπόχνιαρς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι πολύ ικανοποιημένη που άκουσα όλες αυτές τις παρεμβάσεις σήμερα. Η ιδέα της εισαγωγής ποσοστώσεων ασφαλώς δεν είναι ο μοναδικός μηχανισμός. Πρέπει να αναζητήσουμε και άλλους τρόπους για να επιτρέψουμε στις γυναίκες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην πολιτική και να καταλάβουν υψηλέ θέσει. Είμαι πάντως πεπισμένη ότι είναι ο μόνος τρόπος για να επιταχυνθεί η διαδικασία αυτή. Κάτι το οποίο είναι απολύτως αναγκαίο. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Δόκτωρ Κένι Μέριλ. Σας ευχαριστώ για όλες τις ε, τοποθετήσεις σας. Πολλά θέματα προέκυψαν και η αναγκαιότητα να συνδυαστούν διαφορετικές στρατηγικές για να ε, δημιουργηθεί και αυτό το capacity building και θεσμικές ε, αλλαγές, διότι όλοι μιλήσαμε και μιλήσατε και για θεσμούς που έχουν χρειαστεί αιώνε για να δημιουργηθούν και βεβαίως κυριαρχούνται από άνδρες. Σημειώνω και τόσα λέχθηκαν για την ανάγκη να επαγρυπνούμε, διότι όπως πολλές από εσά είπατε, μπορεί να αντιστραφούν τα όσα έχουμε κερδίσει και δεν είναι ε, ε, σίγουρη η πρόοδος. Θα χρειάζεται λοιπόν να παρακολουθούμε διαρκώς την εξέλιξη. Ευχαριστώ πολύ, Δόκτωρ Κένι. Τώρα οι φίλοι μας από την ομάδα των φιλελευθέρων. Κύριε Μλινάρ, θα προσπαθήσω να ε, συνοψίσω σύντομα, αν και σε βάθο. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες και όλους που ήσασταν σήμερα παρούσες και παρόντες σήμερα, και παρόντες εδώ μάλλον, και για τι παρεμβάσει σα. Έχω την εντύπωση ότι ε, είναι κοινό το αίσθημα της ανυπομονησίας. Και εγώ ανυπομονώ. Υπενθυμίζω κάτι που καμιά φορά λησμονούμε. Προερχόμαστε προερχόμαστε, ε, ερχόμαστε μέσα από μια παράδοση ανδροκρατίας χιλιάδων ετών και έχουμε εκλεγεί παρόλα αυτά. Ε, εδώ βρισκόμαστε. Και αυτά βλέπουμε κιόλα τις ημέρες αυτές και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για τα σχόλια ιδίω από την Ιταλίδα συναδελφό μας. Πρώτα για αυτό το... την υπαναχώρηση που βλέπουμε ή την υποχώρηση που βλέπουμε σε ορισμένε χώρε μέλη την αντιμετωπίζουμε και εδώ στο ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή ότι πρέπει να έχουμε πάρα πολύ ξεκαθαρά υπόψη ότι τα πράγματα αυτά δεν είναι γραμμένα στην πέτρα. Και επομένως ε, δεν είναι κάτι που δεν είναι δυνατόν να αντιστραφεί. Άκουσα επίση από την Αυστριακή συναδελφό μου και από τη Λιθουανή συναδελφό μου σημαντικά πράγματα. Όταν λέτε ότι χρειάζεται να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθηση των γυναικών έτσι ώστε να κατέλθουν υποψήφιε, να μπουν στην πολιτική, αλλά και να είναι και βέβαιο ότι δεν θα κολλήσουν εντό εισαγωγικών σε κάποια ελαφρά θέματα, α πούμε, διότι τότε τι παραγωνίζουν και δεν τι λαμβάνουν σοβαρά υπόψη οι άνδρες. Νομίζω ότι όλες το έχουμε ζήσει αυτό. Ήδη η Επιτροπή Δικαιωμάτων Γυναικών δεν είναι νομοθετική επιτροπή. Δεν έχουμε την ίδια νομοθετική βαρύτητα όπως ας πούμε η Επιτροπή Οικονομικών ή Εξωτερικού Εμπορίου. Η σύστασή μου λοιπόν προς όλες τις γυναίκες ε, συναδέλφους είναι προχωρήστε, μπείτε και σε μια από τις σκληρές κοινοβουλευτικέ επιτροπές, αυτές δηλαδή που έχουν ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα. Και να είστε ταυτόχρονα και μέλος της Επιτροπής Δικαιωμάτων Γυναικών. Εγώ είμαι ταυτόχρονα τακτικό μέλο στην Επιτροπή Ενέργεια, Έρευνα και Ενέργεια. Κάτι το οποίο δίνει στο λόγο μου πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα και μέσα στην δική μου κοινοβουλευτική ομάδα, για να μπορώ να προαγάγω και θέματα ισότητα των φύλων. Γιατί εκεί με λαμβάνουν σοβαρά υπόψη οι συναδελφοί μου. Κάτι άλλο το οποίο λέχθηκε και το οποίο πραγματικά θα ήθελα να το λάβετε σοβαρά υπόψη και αναφέρθηκε στην εισαγωγική στην εισαγωγική τοποθέτηση της κυρίας είναι το ζήτημα των συμμαχιών χρειάζεται να φτιάξουμε συμμαχίε. Δεν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για όλα τα πολιτικά θέματα και σε όλου του τομεί. Αλλά μπορούμε να συμφωνήσουμε, α πούμε, στο γεγονό ότι πρέπει να ενισχύσουμε το θεματολόγιο τη ισότητα των φύλων. Χρειαζόμαστε τι συμμαχίε αυτέ. Και κυρίω μην κάνετε το λάθο να θεωρήσετε ότι είναι και διαφορετικά τα πράγματα, διότι η Ευρώπη βασίζεται σε συμβιβασμού και συμμαχίε. Είμαι μεγάλη συνήγορος του συμβιβασμού, διότι εάν όλοι μπορούσαν να συμβαστούν θα ήταν πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα τα πράγματα. Βεβαίω είμαι βεβαία ότι οι δικέ μου ιδέε είναι οι απόλυτα σωστέ, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι αν συμφωνήσουν οι συναδελφοί μου και συμβαστώ μαζί του, θα προχωρήσουν τα πράγματα. Και ιδίω με Ανιέσκα και η Ράτσε που είναι παρούσε εδώ, οι συναδελφοί μου ευρωβουλευτέ, έχουμε συνεργαστεί διακομματικά για θέματα τα οποία μας απασχολούν ιδιαίτερα και έχουμε επιτύχει καλά αποτελέσματα. Λοιπόν, μην το λησμονούμε αυτό. Τώρα, ποσοστώσεις. Α, για μένα που είμαι φιλελεύθερη, οι ποσοστώσεις είναι δύσκολο θέμα να το προβάλλω. Όμως οι φεμινίστριες πάντοτε προβάλλουν ε, τις ποσοστώσεις. Είναι ένας τρόπος για να καταλήξει κανείς κάπου. Όσο δεν έχουμε τα ποσοστά εκπροσωπήσεως που να απηχούν πραγματικά ε, τον αριθμό των γυναικών στον παγκόσμιο πληθυσμό, η ποσοστός είναι ένας τρόπος. Εάν ο όρος ποσόστος είναι το πρόβλημα, πες το αλλιώς, πες το ροσπάνθυρα, ξέρω εγώ. Η Ελληνίδα συνάδελφός μας έδωσε μια ιδιαίτερη οπτική και την ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρέμβασή της. Είπε κάτι πολύ σημαντικό. Χρειάζεται μια στέρεα πολιτική για την ισότητα των φύλων. Αυτό πρέπει να το επεξεργαστούμε και πρέπει να είναι μια μέσο και μακροπρόθεσμη πολιτική. Και ελπίζω το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο που θα εκλεγεί στην 26η Μαΐου να κάνει το θέμα αυτό τέτοιο που να το προωθήσει και να το προωθήσει ισχυρά. Αυτά από την πλευρά μου και για το τελευταίο σχόλιο. Τώρα και εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον Δανέζα συναδελφό μας που μίλησε για ελευθερία, το οποίο είναι κάτι το οποίο ε, αγγίζει πολύ τις πολιτικές μου πεπιθήσεις. Θέλω να τονίσω ότι δημοκρατία χωρίς ισότητα δεν είναι δημοκρατία. Οι γυναίκες πρέπει να είναι ελεύθερες, να ψηφίζουν, να διεξάγουν εκστρατείες, να καταλαμβάνουν θέσεις, να μιλούν εξ ονόματος των κομμάτων τους, ελεύθερες ε, από τοξικές επιθέσεις, από ε, δυσπιστίες κλπ. Αυτά από μένα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ όλες τις ομιλήτρες και όλους όσους πήραν ε, το λόγο. Και η συνάδελφος Γκαρσία Πέρες ε, θα αναλάβει τώρα ως ε, συντονίστρια για το δεύτερο πάνελ. Και σας ζητώ για μία ακόμα φορά συγγνώμη για τη βραχνή μου φωνή. Χθες το βράδυ βράχνες. Please, please, uh, dear friends, take your seats because we have not... Συνάδελφοι, καθίστε σας παρακαλώ γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε τώρα τη συζήτηση έτσι ώστε να δώσουμε σε όλες σας και όλους τη δυνατότητα να πάρουν το λόγο. Οπότε πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα, άμεσα. I will take uh, the floor in Spanish. Maybe you... Please. Θα περάσω στα ισπανικά, ίσως χρειάζεται, χρειάζεται τα ακουστικά σας. Καλημέρα σας σε όλες. Ξεκινάμε το δεύτερο πάνελ που αφορά τη συμμετοχή των νέων γυναικών στην πολιτική. Και για αυτή τη συζήτηση έχουμε μαζί μας δύο μιλήτριες, τις οποίες ευχαριστώ γιατί θέλησαν να συμμετάσχουν σε αυτή τη συνάντηση. Η συντρόφισσά μου η Ινές, η οποία ήταν και ευρωβουλευτής και έχουμε συζητήσει στο παρελθόν μαζί της. Σας ευχαριστώ και όλες εσάς που είστε παρούσες. Είμαστε το 52% της Ευρώπης. 52% στην Ευρώπη είναι γυναίκες. Εάν οι γυναίκες δεν στηρίξουμε τις άλλες γυναίκες, δεν υπάρχει ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Δεν μπορούμε οικοδομήσουμε τις χώρες μας. Δεν μπορούμε να στήσουμε τις πόλεις μας. Γι' αυτό η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική είναι θεμελιώδες στοιχείο. Επιτρέψτε μου να θέσω δύο πράγματα και θα δώσω αμέσως μετά το λόγο στις ε, ομιλήτριές που είναι εδώ. Θα ήθελα αυτό το χρόνο να τον χρησιμοποιήσω για δύο μικρούς προβληματισμούς, για δύο μικρές σκέψεις. Πρώτον, η Ευρώπη είναι ένα οικοδόμημα που στηρίζεται σε αξίες και μεταξύ αυτών των αξιών βρίσκεται η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Εκείνες που συμμετέχουμε και πιστεύουμε στην Ευρώπη έχουμε την ευθύνη και την υποχρέωση να υλοποιήσουμε αυτές τις αξίες, να προωθήσουμε την ισότητα. Δεν είναι τυχαίο που παίρνουμε αυτές τις αποφάσεις. Δεν είναι τυχαίο όπου υπάρχουν κυβερνήσεις που δεν υπάρχει ούτε μία γυναίκα. Δεν είναι τυχαίο που οι δείκτες συμμετοχής των γυναικών στα εθνικά κοινοβούλια είναι κάτω από τα ποσοστά των ανδρών. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά τα πράγματα. Είναι η ίδια η Ευρώπη η οποία έχει άνισες δομές. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσπαθήσουμε, πρέπει να δεσμευτούμε, άντρες και γυναίκες, όσοι πιστεύουμε στην ισότητα, ως βασικού άξονα της πολιτικής μας πρέπει να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Για να γίνει αυτό πραγματικότητα, οι ποσοστώσεις είναι βασικό εργαλείο και μας βοήθησε και εμάς πολλές από τις γυναίκες πολιτικούς για να φτάσουμε εδώ. Χωρί αυτέ τι ποσοστώσει δεν θα είχαν φτάσει οι γυναίκε σε αυτέ τι θέσει για να λαμβάνουν μαζί με του άντρε αποφάσει. Χάρη σε αυτέ τι γυναίκε. χάρη στι φεμινίστριες που δούλεψαν στις προηγούμενε γενιές πριν φτάσουμε εμεί εδώ, εμεί φτάσαμε σε αυτέ τι θέσει. Θα ήθελα λοιπόν να χρησιμοποιήσω αυτό το χώρο και αυτό το χρόνο για να ευχαριστήσω όλε εκείνε τι φεμινίστριες που έφτιαξαν κοινωνίε πιο ίσε, πιο δίκαιε. Και εμείς είμαστε σήμερα εδώ διεκδικώντας ξανά τα δικαιώματά μας. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε οι κόρες μας να έχουν λιγότερα δικαιώματα από εμά, τις μητέρες. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε ένα μεγάλο καθήκον να υλοποιήσουμε, να υλοποιήσουμε αυτή την ισότητα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να βροντίξει η μία λέξη στους δρόμους της Ευρώπης μία κραυγή, κραυγή της ισότητας, για να φτιάξουμε την Ευρώπη που όλοι θέλουμε. Και τώρα, μετά από αυτά τα λίγα λόγια, θα δώσω το λόγο στη συντρόφισά μου και φίλη μου, Ανέ Στούμπερ, μέλος του Δημοκρατικού Κινήματος Γυναικών της Πορτογαλίας. Ήταν συντροφός μου στην Επιτροπή Γυναικών εδώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για κάποια χρόνια και για μένα είναι μεγάλη χαρά που τη δίνω τώρα το λόγο για να πει και αυτή τι δικές της σκέψεις σε αυτή την εκδήλωση. Ινέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω στα πορτογαλικά. Ευχαριστώ, Ράτσε. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω ε, για αυτή την πρόσκληση από την πλευρά τη Επιτροπή. FM. Εγώ ε, θα σας θα δώσω μια έμφαση σε μια διαφορετική οπτική γωνία και στο ε, ε, γεγονός ότι η αύξηση των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών έχει να κάνει με την πιστοδρόμηση σε ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας και τις οικονομικές συνθήκες ε, των γυναικών. Έχουμε δηλαδή εδώ οικονομικού, κοινωνικού και πολιτισμικού χαρακτήρα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας. Δηλαδή μιλάμε για προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλε οι γυναίκε, αλλά ειδικότερα οι γυναίκε χαμηλότερου εισοδήματος. Ε, δηλαδή δεν μπορούμε να ε, συζητούμε το ζήτημα των διψενών διακρίσεων χωρί να εξετάζουμε την οικονομική κατάσταση και την κοινωνική προέλευση ε, των γυναικών. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση ουσιαστικά βρισκόμαστε όλο ένα και πιο μακριά από το να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτέ τι γυναίκε να συμμετάσχουν στην πολιτική και γενικότερα στα, στα κοινά. Δηλαδή οι, αυτές η, η, αυτή η κατάσταση οδηγεί στις διάφορες δυσμενεί ει ε, των γυναικών ε, ε, πρακτικές ε, θα ήθελα να σα δώσω κάποια παραδείγματα σε ό,τι αφορά τους πραγματικούς λόγου, πραγματικές αιτίε, οι οποίες εμποδίζουν τις γυναίκες από το να συμμετάσχουν στην πολιτική ζωή. Και εδώ για παράδειγμα έχουμε την αύξηση της επισφαλούς και της μερικής ε, αργασίας, η ε, επιβολή ουσιαστικά κυρώσεων ε, σε ό,τι αφορά την μητρότητα, η ανυπαρξία μηχανισμών κοινωνικής υποστήριξης και ό,τι καθεξής. Να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Η αύξηση της εργασιακής εκμετάλλευσης και της επισφαλούς εργασίας είναι, αφορά περισσότερο τις γυναίκες για παράδειγμα, ε, το 1 τρίτο των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζονται με αυτέ τι συνθήκε. Στη δική μου χώρα το 21,5% το 2013 των γυναικών ε, που εργάζονταν δεν είχαν ε, σύμβαση αορίστου εργασία και το 60% από αυτέ ήταν το 60% στις γυναίκες κάτω των 25 ετών βρίσκονταν σε αυτή την κατάσταση και το 33% των γυναικών 25 και 30, από 25 έως 34 ετών. Και βέβαια η μερική εργασία και αυτή ε, έχει να κάνει περισσότερο με γυναίκε. Δηλαδή ε, το 2013 64% των γυναικών στη δική μου χώρα ε, εργαζόταν σε βάρδιε, σε τη νύχτα, τα Σάββατα ή τι Κυριακέ. και γι' αυτό βέβαια έχουμε αντίστοιχα δηλαδή με αυτή την υπερεκπροσώπηση στη μερική και επισφαλή εργασία των γυναικών και χαμηλότερε αποδοχέ για τι γυναίκε. Δηλαδή το μισθολογικό χάσμα μεταξύ άνθρωπων και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο 16%. Εάν Λοιπόν, εγώ είμαι μια γυναίκα που ε, λαμβάνει το κατώτατο μισθό των 600 ευρώ στην Πορτογαλία. Θα πρέπει να δω κατά πόσο θα καταφέρω να επιβιώσω στο τέλο του μήνα ε, πληρώνοντα του λογαριασμού ε, μου και να δω ε, από εκεί και μετά όταν θα τελειώσει η εργασιακή μου σύμβαση πώ θα βρω νέα εργασία. Ενώ θα πρέπει να προσαρμοστώ στο να ε, μία εβδομάδα να εργάζομαι τη νύχτα ή την επόμενη εβδομάδα να εργάζομαι ε, το Σαββατοκύριακο και να δω πώ μπορώ να, να ανταποκριθώ σε όλε τι υποχρεώσει που έχω και σε οικογενειακό επίπεδο αν έχω ανήλικο παιδί. Άρα λοιπόν υπό αυτή την κατάσταση έχω τη δυνατότητα, έχω ε, την, την πολυτέλεια αν θέλετε να συμμετάσχω στην πολιτική ζωή, δεν το νομίζω. Ε, άρα λοιπόν παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μου λέει ότι θέλει να έχω περισσότερη ε, εκπροσώπηση στην πολιτική ζωή, ε, θα πρέπει αντιθέτω να, να μου προσφέρει περισσότερη εργασιακή ευελιξία. Ένα δεύτερο ε, παράδειγμα είναι ε, το ζήτημα της ε, μητρότητας. Ε, δηλαδή χρειάζεται να αυξήσουμε τη σχετική περίοδο που προβλέπεται στην οδηγία γιατί η ισότητα σε ό,τι αφορά τον μισθό επηρεάζεται από, το να, από την υποχρέωση ουσιαστικά του ο πατέρα, να πρέπει και αυτό να πάρει την άδεια πατρότητα. γιατί ε, χωρίς να υπάρξει διαφοροποίηση ουσιαστικά το να επιβάλλουμε αυτή τη λήψη τη άδεια από τον πατέρα σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε χαμηλότερες αποδοχές για μια οικογένεια. Άρα λοιπόν θα πρέπει να διασφαλίζουμε και την ε, χορήγηση αυτή τη άδεια και αποζημίωση 100% έτσι ώστε και οι γυναίκες να έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να μπορούν να συνεχίσουν την εργασιακή του ε, ζωή και να ε, έχουν τα δικαιώματα μετρότητα, χωρίς δηλαδή να υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις για αυτές. Τώρα, ένα τρίτο παράδειγμα είναι η πρόσβαση στο κοινωνικό δίκτυο των ε, υπηρεσιών φροντίδα. Το σχετική έκθεση που έγινε σε ό,τι αφορά την ισότητα των δύο φύλων του 2014 2015 έφτανε στο συμπέρασμα ότι οι περικοπές που έγιναν στις ε, κοινωνικέ παροχέ, ειδικότερα στη δημόσια υγεία και ούτω καθεξής, βοήθησε στο να περάσει αυτή η ευθύνη, αν θέλετε, για την παροχή αυτών των υπηρεσιών στο ιδιωτικό τομέα και κυριότερα από τις ε, γυναίκες. Όπως αναφέρεται στην έκθεση ε, δηλαδή, υπάρχουν προβλήματα ε, σε ό,τι αφορά, ε, για παράδειγμα, την ε, παροχή και υπηρεσιών σε ό,τι αφορά τη φροντίδα των παιδιών ηλικιωμένων και αυτό έχει βέβαια και ω αποτέλεσμα το να μην συμμετέχουν στην εργασιακή ζωή οι γυναίκε ή μόνο μερικώ. Για παράδειγμα, το 2015 το 29% των γυναικών μεταξύ 20 και 64 ετών δεν ήταν ενεργέ εργασιακά. Εάν λοιπόν εγώ είμαι μια γυναίκα η οποία ε, ε, ε, κερδίζει μόνο 600 ευρώ το μήνα το, το ελάχιστο μισθό και θα πρέπει να δίνω 300 ευρώ από αυτά για, να, για ένα βελφονιπιακό σταθμό, προφανώς μάλλον δεν θα επιλέξω να εργάζομαι. Και αν έχω από εκεί και μετά και έναν ηλικιωμένο συγγενή τον οποίο πρέπει να φροντίζω, δεν έχω καν την επιλογή. Είμαι αναγκασμένη να μην εργάζομαι. Άρα λοιπόν... Αυτέ είναι οι καταστάσει οικονομικές οι οποίες ε, παίζουν αποφασιστικό ρόλο και θα πρέπει να διασφαλίσουμε τις ελάχιστες ε, προϋποθέσεις για όλες τις ε, γυναίκε. Εάν δούμε τώρα την σύνθεση των εκλογικών ληστών και του διορισμού στις διάφορες δημόσιες επιχειρήσεις βλέπουμε ότι πάντοτε ξεχνάμε ε, την μεγάλη πλειοψηφία των γυναικών. Ε, δηλαδή, ε, προφανώ θέλουμε να υπάρχει εκπροσώπηση των γυναικών, αλλά αν εστιάσουμε μόνο εκεί, δηλαδή στι ε, πολιτικέ λίστε, στι ε, υψηλέ θέσει, τότε θα ξεχάσουμε τη μεγάλη ε, πλειοψηφία των γυναικών, ειδικότερα εκείνων οι οποίε βρίσκονται στα χαμηλότερα κοινωνικά ε, στρώματα. με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, θα υπερασπίσουμε την, τα, τα, δικαιώματα τη ε, συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών. Και μάλιστα έχουμε δει ότι και εκείνε οι γυναίκε που βρίσκονται σε υψηλό αυτές ε, δεν ε, έχουν σταματήσει την, τις αποφάσεις που ε, έλαβαν. Δηλαδή το γεγονός ότι ορισμένες επίτροποι, ορισμένες γυναίκες σε πολιτική ήταν σε αυτές τις θέσεις και ήταν γυναίκες δεν τους παρεμπόδισε από το να λάβουν αποφάσεις οι οποίες οδήγησαν σε επαναχώρηση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε ε, μια ε, νέα προσέγγιση με βάση την οποία όλες οι γυναίκε θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ε, ζωή και δεν θα πρέπει αντιθέτω να δημιουργήσουμε μια τεχνητή εντός εισαγωγικών ισότητα και από εκεί και μετά εμείς από το κίνημα της μάλλον σήμερα σε μια ε, στη σημερινή Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας ε, από την πλευρά του ε, Δημοκρατικού Κινήματος για τις Γυναίκες οργανώνουμε και μια διαδήλωση προκειμένου για, τρίτο συνεχόμενο έτος ώστε να συνεχίσουμε τον αγώνα που δίνουμε για πιο ισόρροπη εκπροσώπηση των γυναικών. Ευχαριστώ πολύ, Ινές. Θα περάσουμε κατευθείαν στην επόμενη ομιλήτρια. Καρίμα Ζαΐ, που είναι μάνατζερ της εκστρατείας ε, Equal Brussels για τη δημόσια διοίκηση της περιφέρειας των Βρυξελών. Θα μας παρουσιάσει θέματα πολύ σημαντικά για τη δουλειά μας και τον αγώνα μας. Ευχαριστώ, Ιράτσε. Θα μιλήσω αγγλικά. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν εκπροσωπώ σήμερα την ε, περιφέρεια των Βρυξελών και τη δημόσια διοίκησή της. Παρότι έχω δουλέψει ως campaign manager εκεί, ε, κάναμε μια εκστρατεία για την ε, σεξουαλική βία στην περιφέρεια των Βρυξελών. Ίσως απογοητευτείτε που δεν βλέπετε μια νέα γυναίκα να μιλάει, κι όμως είμαι νέα γυναίκα. Αλλά δεν είμαι εδώ για να εκπροσωπήσω και να μιλήσω εκ μέρου των νέων γυναικών. Θέλω να σας μιλήσω για την εμπειρία μου. Για ένα θέμα που μίλησαν και στο προηγούμενο πάνελ ε, που αφορά τις γυναίκες στην πολιτική, την εξουσία των ε, γυναικών πολιτικών. Και πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε την ισότητα ανδρών και γυναικών στην πολιτική. Χρειάζεται και Ποιοτική συνεισφορά βέβαια. Συμφωνώ με τα όσα είπε η κυρία Κένι Μέριλ. ότι πρέπει να τις βοηθήσουμε τις γυναίκες για να καταλάβουν το πρόβλημα της υποεκπροσώπησης. Δεν το έχουν οι ίδιες. Εμείς ε, κάναμε ένα πρόγραμμα για τις μετανάστριες γυναίκες όπου συμμετείχαν διάφορα πολιτικά κόμματα. Από τις προηγούμενες εκλογές δούλεψα για το λόμπι των Ευρωπαίων γυναικών και συντόνισα την, το πρώτο δίκτυο για το mentoring των γυναικών που ξεκίνησε το, στις 9 Απριλίου του 2013 ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Αυτό το πρόγραμμα ε, ήταν τμήμα ε, του πλαισίου μια, που προωθούσε μια εκστρατεία 50-50, 50%, 50 άντρες, 50% αντρες 50 γυναικες Με σκοπό την, εκπροσώπηση, την καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ε, και το να συζητηθούν θέματα για, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ισότητα των φύλων και να μπουν ψηλά στην ατζέντα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Είναι ένα από τα πρώτα δίκτυα τέτοιας φύσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σε εξηγήσω περί την επρόκειτο. Είχαμε 11 γυναίκες ευρωβουλευτές που ενδιαφερόταν να κατέβουν σε εκλογές του 2014, τις ευρωεκλογές εκείνες. Για να τις προετοιμάσουμε, θέλαμε να τις προετοιμάσουμε και να τις στηρίξουμε μέσω του δικτύου ε, καλύτερα για να έχουν περισσότερες ευκαιρίες. Μία από τη Σλοβενία, από τους σοσιαλιστές, η Μόικα Σοβίνια, η Ούλικα από τους ε, πράσινους της Αυστρίας. Ήταν δύο από τι γυναίκες. Θέλαμε να ενισχύσουμε τις δεξιότητες, την αυτοπεποίθηση και τη δικτύωση αυτών των νέων γυναικών και να τις εξοπλίσουμε καλύτερα ε, ως υποψήφιες ε, ευρωβουλευτίνες. Ε, αντάλλαξαν εμπειρίες στις συνεδριάσεις με το μέντορά του, συμμετείχαν σε διασκέψεις, σε συνεδριάσεις, για τη δημοκρατία μέσα στα κόμματα και σε αυτή την αίθουσα μάλιστα ετοιμάσαμε μια εκδήλωση ε, με τίτλο «Ο Ευρωβουλευτής μου είναι σαν και εμένα». Ε, γιατί προσπαθούσαμε να βρούμε ανθρώπους με τα οποία θα ταυτίζεται ο Ευρωπαίος ψηφοφόρος. Ε, επίσης, μια γυναίκα, η Λίντα Κόεν, είπε ότι αν οι γυναίκες δεν κάθονται στο τραπέζι που λαμβάνονται τις αποφάσεις, τότε θα βγουν και από το μενού. Αυτό μου μείνε. Και δυστυχώς ισχύει ακόμα και σήμερα. Άλλα πράγματα που θεωρούσαμε σημαντικά είναι να δημιουργηθούν δίκτυα, γιατί έλειπε αυτό από τις γυναίκες οι οποίες μπαίνουν στο στίγμα της πολιτικής. Το πρόγραμμα μιλούσε για την ηγεσία, και την αύξηση του δυναμικού, ε, την ε, αύξηση των γνώσεων για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και την επικοινωνία. Συζητήσαμε τότε και είναι σημαντικό και σήμερα το πώς θα αποκτήσουν δεξιότητες για να αντικρούσουν δημαγωγικά επιχειρήματα, λαϊκιστικά επιχειρήματα και να χρησιμοποιήσουν και να καταλάβουν μάλλον τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι λαϊκιστές για να μπορέσουν να μιλήσουν πιο πιστικά στους εκλογείς του, στο εκλογικό σώμα. Ε, υπάρχει ένα κίνημα ε, αυτή τη στιγμή κατά τη ισότητα των φύλων και ακριβώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, το καταπολεμήσουμε με αυτά τα όπλα. Επίσης, χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, τις βοηθήσαμε να συμμετέχουν σε διάφορες συνεδριάσεις επιτροπών, ολομέλειας κτλ. Να παρακολουθήσουν δηλαδή τις εργασίες του Κοινοβουλίου. Εκείνη την εποχή διάφορες ε, γυναίκες πολιτικές ε, συνήλθαν, ε, κατοντάδες γυναίκες από διάφορα κοινοβούλια για να συνειδητοποιήσουν το ρόλο τους στην πολιτική. Είναι σημαντικό να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις γιατί χρειαζόμαστε και μοντέλα αλλά οι γυναίκες χρειάζονται να πλαισιώνται από άλλες γυναίκες που έχουν ήδη καταλάβει υψηλά αξιώματα για να εμπνέονται από εκείνε. Η μοναδικότητα αυτού του προγράμματός μας ήταν ότι είχε μια ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία. Ε, χρηματοδοτήθηκε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, το δημόσιο αυτό χρήμα ξοδεύτηκε καλά. Ε, Ήθελα να τις φέρει πιο κοντά στην, στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Οι μέντορες προσπαθούσαν να τις βοηθήσουν να αυξήσουν το δυναμικό τους, γιατί αυτές οι γυναίκες είναι πολίτες και χάρη στην πολιτική τους δραστηριότητα θα μπορούσαν να βοηθήσουν άλλους να αποκτήσουν δύναμη. Ένα παράδειγμα είναι μια γυναίκα που εξελέγει πρόσφατα η πρώτη δήμαρχος της Καραϊβικής, μιας πόλης της Ήταν υποψήφια στις τελευταίες ευρωεκλογές, αλλά δεν ήταν ψηλά στον εκλογικό κατάλογο των, των σοσιαλιστών. Επίσης υπάρχει μια άλλη ε, υποψήφια των Πρασίνων στην Ολλανδία, ε, υποψήφια στις τελευταίες εκλογές. Καταλήγοντας, το πρόγραμμα αυτό δημιούργησε έτσι μια συνειδητοποίηση ε, για το θέμα της ισότητας και ειδικά για τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι νέες γυναίκες έχρωμες, ε, οι οποίες ενδιαφέρονται να κατέβουν στην πολιτική. Είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αντανακλά την ποικιλομορφία όλων των ευρωπαϊκών λαών είναι σημαντικό να υπάρχει ισότητα των φύλων, που είναι και το σημαντικό μας θέμα σήμερα, αλλά να υπάρχει εκπροσώπηση και όλων των ηλικιών, ε, της εθνικής προέλευσης και όπως είπε η Νές, να λάβουμε υπόψη μας την ποικιλομορφία. Οι γυναίκες από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα να εκπροσωπούνται επίσης. Πολύ συχνά αντιμετωπίζουμε νεποτισμό, ε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολλαπλά αξιώματα, ένας άνθρωπος πολλά αξιώματα. Τι πράγμα... Αυτή η νοοτροπία είναι μολυσματική. Δεν είναι κληρονομική αρρώστια, αλλά είναι μεταδοτική θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ισότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε εθνικό επίπεδο φυσικά, γιατί υπάρχει ένα σύνδεσμο ανάμεσα στα δύο επίπεδα. Πρέπει η ισότητα να επιτευχθεί καταρχά σε επίπεδο κράτου μέλου. Είναι σημαντικό να υπάρχουν και θετικά μέτρα δράση για να έρθουμε κοντά σε αυτέ τι γυναίκε σε εθνικό επίπεδο, και να δούμε ποιε είναι οι γυναίκε που έχουν το δυναμικό, που έχουν τα φόντα να μπουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τώρα πραγματικά τελειώνω. Ένα μεγάλο μοντέλο, ε, ένα μεγάλο πρότυπο ε, για τους πολιτικούς είναι η κυρία μέλο ε, μέλος Παγκόσμιας Τάπεζας, που είπε ότι και η ίδια θεωρούσε ότι το να, το να αποκτήσει κανείς αυτοπεποίθηση είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, ήταν σημαντικό στοιχείο και για την ίδια. Και κάθε φορά που άνοιγε ένα υψηλό πόστο, αμφέβαλε για το κατά πόσο θα μπορούσε να το πάρει, αν το και αν είχε τα προσόντα για να το πάρει. Και είπε ότι κανένας θεσμός, καμία χώρα δεν μπορεί να τα καταφέρει εάν δεν αξιοποιήσει το δυναμικό όλων των ανθρώπων που έχει, ανδρών και γυναικών. Ευχαριστώ και τις δύο μιλήτριες και τώρα θα γίνει μια συζήτηση. Υπάρχουν διάφοροι που ζήτησαν το λόγο, όπως και στο προηγούμενο πάνελ. Ξέρετε ότι ο καθένας έχει πάνω κάτω δύο λεπτά. Το κάνουμε αυτό για να έχουμε το, τη δυνατότητα να δώσουμε το λόγο σε όλους όσους το επιθυμούν και για να μπορέσουν και οι δύο μιλήτριες να σας απαντήσουν και να τελειώσουμε βεβαίως εν καιρός. Η κυρία Ρωμάνα Χέροβικ από την Κροατία έχει το λόγο. Μπορεί να το πρόφερα τόσο άσχημα το όνομα που δεν καταλάβατε ότι είστε εσεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έδωσα το όνομα σε αυτήν την κυρία από την Κροατία. Μπορεί να μην κατάλαβε καν το όνομά τη, όπω το πρόφερα, βέβαια. Ζητώ συγγνώμη, γι' αυτό ξαναπέρνω το λόγο. Σίγουρα σας ε, σκότωσα το όνομά σας. Α, δεν είναι εδώ αυτή η κυρία. Πάμε στην επόμενη, η κυρία Κριστίνα Γιουρισνίτη από την Ρουμανία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω γαλλικά εγώ. Είμαι υπέρ της ισότητας των φίλων αλλά και των γλωσσών. Και θα μιλήσω υπό την ιδιότητα της εκπαιδευτικού γιατί είμαι καθηγήτρια γαλλικών και θα ήθελα να απαντήσω στην ε, Ινιές, να πω δηλαδή ότι είναι αλήθεια ότι αν δεν έχει κανείς χρόνο, αν έχει παιδιά, αν έχει δυσκολίες στο επάγγελμα, είναι πολύ δύσκολο να μπει κανείς στην πολιτική. Δεν έχει δηλαδή επαρκή χρόνο μια γυναίκα για να γίνει πολιτικός και να μπορέσει να στρατευθεί, ε, να διαθέσει ενέργεια και να αναλάβει ευθύνες. Είναι πολύ δύσκολο και εγώ ίδια είμαι η γυναίκα, μεγαλώνω μόνη το παιδί μου, ε, έχω μεγάλες δυσκολίες να μπορέσω να αφιερωθώ στην πολιτική πέρα από τα καθημερινά προβλήματα. Μπόρεσα να αναμειχθώ στην πολιτική εδώ και δυόμιση χρόνια, διότι ο γιος μου είναι πια ενήλικος, έχει αρχίσει να δουλεύει, ε, άρα έχω μια ελευθερία. Άρα είναι σωστό, οι γυναίκες έχουν δυσκολία να εμπλακούν στην πολιτική, διότι έχουν ας πούμε τα οικιακά, τα ψώνια, έχουν ε, να μεγαλώσουν τα παιδιά, που είναι τα πρώτη στα καθήκοντα για τις γυναίκες. Δεν υπάρχει διέξοδος. Ως εκπαιδευτικός μπορώ ωστόσο να σας πω με σαφήνεια ότι τα θετικά μέτρα για τα οποία μιλήσαμε σήμερα δεν μπορούν να εφαρμοστούν αν δεν υπάρχει ένα υπόβαθρο παιδείας. Διότι κάθε εξέλιξη βασίζεται στην παιδεία. Δυστυχώς η Ρουμανία δεν έχει ποιοτικά προγράμματα ανταλλαγών. Τα, ε, τα προγράμματα των σχολών είναι γεμάτα από στερεότυπα και για τα φύλλα και για τα γενετήσια δικαιώματα και αυτά στο 90% των σχολείων. Σε ό,τι αφορά τη δραστηριότητά μου έως τώρα ως βουλευτού, εγώ έχω ρίξει ιδιαίτερο βάρος στην παιδεία και για θέματα ε, ισότητας φύλου αλλά και σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Έχω οργανώσει σεμινάρια, εργαστήρια, ε, δημόσιες συναθρήσεις για τα θέματα αυτά και έχω αναλάβει και νομοθετικές πρωτοβουλίες στο επίπεδο του Ρουμανικού Κοινοβουλίου. Ψηφίσαμε μεν ε, πρόσφατα για να μπούμε και στην ε, σύμβαση της ε, Κωνσταντινούπολης και την κύρωση Ρουμανία το 2016 μαζί με αυτά και τα υποχρεωτικά για την παιδεία, ωστόσο δεν έχει επέλθει καμιά αλλαγή και δεν προβλέπεται καμιά αλλαγή για το επόμενο σχολικό έτος. Άρα στο επίπεδο της παιδείας έχουμε σημαντικές δυσκολίες για να προδέσουμε. Άρα πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά πράγματα. Πρέπει να συνεχίσει κανείς τον αγώνα όμως και να έχει και πεποίθηση. Εύχομαι σε όλες τις γυναίκες που είναι σήμερα παρούσες εδώ καλή τύχη, καλή δουλειά και καλή ε, επιτυχία σε όσα επιθυμούν. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαρία Λαριστίδου από την Κύπρο. Καλή σας μέρα. Εάν τα εμπόδια που συναντούν οι γυναίκε για πρόσβαση στην πολιτική είναι μεγάλα, τα εμπόδια που συναντούν οι νεαρέ γυναίκε είναι σχεδόν ανυπέρβλητα. Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, οι Κύπριες γυναίκες αντιμετωπίζουν εμπόδια που δυσχεραίνουν την ενασχόλησή τους με την πολιτική. Οι πολιτισμικές στάσεις ως προς το κοινωνικό ρόλο των γυναικών υπερτονίζουν τον αναπαραγωγικό και μητρικό τους ρόλο, παρεμποδίζοντας τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η ύπαρξη ποιοτικών και οικονομικά προσιτών δομών παροχής φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων εκτιμάται ότι θα συντελέσει στη διευκόλυνση της εμπλοκής των γυναικών στην πολιτική. Το κυρίαρχο αντρικό μοντέλο άσκησης εξουσίας, το οποίο στηρίζεται στις παραδοσιακές στάσεις περι... των γυναικών από την πολιτική, εμποδίζει την ισόρροπη αντιπρόσωπευση των γυναικών στην πολιτική ζωή και τα πολιτικά κόμματα. Θετικά μέτρα τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην αλλαγή της κυρίαρχης κουλτούρας στα πολιτικά συστήματα είναι η διευκόλυνση της συμφιλίωσης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, η οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών, η υιοθέτηση μέτρων για ενίσχυση των ηγετικών ικανοτήτων των γυναικών, η θετική προβολή της εικόνας των γυναικών από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η ανατροπή των έφυλων στερεοτύπων και των παραδοσιακών αντιλήψεων με βάση το κοινωνικό φύλλο στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών συστημάτων. Συγκεκριμένε πρωτοβουλίε απαιτούνται επίση για την ενδυνάμωση των γυναικών, για υποβολή υποψηφιότητα ποιότητας συμπεριλαμβανομένη της δικτύωσης, της καθοδήγησης και της ανάπτυξη δεξιοτήτων. Οι κοινοβουλευτικοί μπορούν να διαδραματίσουν καταλητικό ρόλο στην προώθηση της ισόρροπη συμμετοχή των δύο φύλων στην πολιτική μέσω τη άσκηση αποτελεσματικότερου ελέγχου επί του αντιχτύπου της νομοθεσίας στα δύο φύλλα ξεχωριστά και επί των δράσεων τη εκτελεστική εξουσία. Κλείνοντα όμω, θα ήθελα να αναφερθώ και σε ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, ειδικά για το πολιτικό μέλλον των νεαρών γυναικών στην πατρίδα μα. Αυτών δηλαδή που επιθυμούν να εμπλακούν ενεργά και στην πολιτική ζωή. Πιστεύω ότι ο κυπριακό λαό έχει οριμάσει και δεν διακατέχεται από αγκυλώσει του παρελθόντο, όπου η εκτίμηση του για τη γυναίκα ήταν περιορισμένη. Σήμερα έχουν αλλάξει προ το θετικό όλα αυτά, λαμβάνοντα μάλιστα υπόψη ότι στι τελευταίε βουλευτικέ εκλογέ είχαμε κάπω αυξημένη εκπροσώπηση ε, των γυναικών στη Βουλή και μάλιστα σε νεαρή ηλικία μεταξύ των οποίων και υποφαινόμενοι. Πιστεύω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και ελπίζω να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή ε, στη συνέχεια και μόνο ενωμένε μπορούμε να αγωνιστούμε για μια καλύτερη κοινωνία και για τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών. Σας ευχαριστώ. Thank you, Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ μέλος τώρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κυρία Κούνεβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χρόνια πολλά και αγωνιστικά σε όσες και όσους στηρίζουν τις γυναίκες, την ισότητα των φίλων και μάχονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νέες γυναίκες και πολιτικοί. Γιατί όμως το συζητάμε, τα αναρωτηθεί κανείς, δεν υπάρχουν τόσα δικαιώματα γυναικών που καταπατούνται καθημερινά. Γιατί δεν συζητάμε για τους κινδύνους φτωχοποίησης των νέων γυναικών, οι οποίοι είναι περισσότερα από ό,τι για τους άντρες. Γιατί δεν μιλάμε για τα εμπόδια που μετά από χρόνια συζητήσεων εξακολουθούν εφίστανται στην αγορά εργασία για τις γυναίκες, για τις ανισότητες μισθούς σε συντάξεις γιατί δεν μιλάμε για τη βία ενάντια στις γυναίκες, γιατί χρειάζεται πολιτικές και μέτρα που θα δώσουν λύσεις στα προβλήματα αυτά. Συζητάμε για τις νέες γυναίκες και την πολιτική όχι μόνο γιατί έρχονται οι ευρωεκλογέ και θα πρέπει να μειωθούν οι ανισότητες που υπάρχουν ως προς την εκπροσώπηση των φίλων στην πολιτική σκηνή, αλλά κυρίως γιατί σήμερα έχουμε και πάλι την ανάγκη να αναδείξουμε την φεμινιστική πολιτική ψηλά στην ατζέντα, γιατί εδώ και καιρό τα ανθρώπινα δικαιώματα και κατά συνέπεια τα δικαιώματα των νέων γυναικών έχουν αντικατασταθεί από τα οικονομικά, τραπεζικά, νομισματικά δικαιώματα, όχι όμως των πολιτών, αλλά των συστημικών θεσμών. Χρειαζόμαστε νέες γυναίκες στην πολιτική, αλλά γιατί γιατί θα συνεισφέρουν κάτι διαφορετικό, γιατί θα συνεισφέρουν κάτι παραπάνω. Δεν θα το μάθουμε αν δεν υπάρξουν οι συνθήκες που θα τους επιτρέψουν να συνεισφέρουν ό,τι μπορούν. Γιατί μέχρι σήμερα, από το 1979, που ξεκίνησε η λειτουργία της Επιτροπής Γυναικών ως Εξατιστικής Επιτροπής, ξέρετε πόσες οδηγίες και θέματα ισότητας πέρασαν περίπου 10. Μέσα λοιπόν σε περίπου 40 χρόνια, μόλις 10 νομοτεθήματα, Μα γιατί πάμε με ρυθμούς χελώνας. Μια από τις απαντήσεις τις βρίσκεις εύκολα αρκεί να δεις την κατανομή των θέσεων των προηγούμενων κοινοβουλίων, των κολέγιων, των επιτροπών, των επικεφαλής των κρατών μελών. Φταίνε οι άντρες, θα ρωτήσει κανείς. Φταίνε οι ανισότητες, θα σας απαντήσω. Και από αυτές κουβαλάμε όλα τα φύλλα. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε νομοθετήματα που να βοηθούν τα φύλλα να έρθουν πιο κοντά σε μια πραγματική ισότητα. Δεν ξέρω αν το, θα το πετύχουμε αυτό με το τελευταίο μας κείμενο την οδηγία για την προσωπική και επαγγελματική ζωή. Προσωπικά πολύ φοβάμαι έχοντας δει το τελικό κειμένο μετά τους τριλόγους. Αμφιβάλλω ότι ακόμα και αν το επόμενο κοινοβούλιο αποτελείται από ίσο ρυθμό γυναικών και ανδρών, καταφέρει να επιφέρει την ισότητα στην Ένωση. Δεν μπορεί να έρθει αλλαγή μαγικά. Υπάρχουν οι συνθήκες που διονίζουν τα στερεότυπα, που βάζουν εμπόδια που περιορίζουν. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν. Πολιτικές που να επελευθερώνουν την γυναίκα από τα εμπόδια, από τα στερεότυπα, από το πατριωτισμό, πατριαρχισμό. Συνάδελφοι, καιρός να επελευθερωθούμε από τα στερεότυπα που ακολουθούν τα φύλλα. Δεν νομίζετε. Αν ναι, τότε θα συμφωνήσετε με την φράση της Ρόζα Λουξεμπουργκ. Η ελευθερία των κοινικών σημαίνει κοινωνική ελευθερία. Αν δεν σας αρέσει να λέτε πως είστε φεμινίστρες, δεν πειράζει. Αρκεί να μάχεστε για κοινωνική ελευθερία. Αυτή θα φέρει και την ελευθερία των κοινικών. Σε ευχαριστώ. Thank you, Mrs. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κούνεβα. Ακολουθεί η κυρία Μαρία Κελερέτη από την Ελλάδα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα συμφωνήσω και εγώ με την εισηγήτρια από την Πορτογαλία και θέλω με τη σειρά μου να επισημάνω ότι η απορρίθμιση στην αγορά εργασίας, η επισφάλεια στην εργασία, οι ευέλικτες μορφές εργασίας ε, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί με την κρίση και τις πολιτικές λιτότητας, είναι ένα από τα βασικά εμπόδια των νέων γυναικών να μπορούν να συμμετέχουν ε, στην πολιτική ζωή. Ο καθημερινός αγώνας για την επιβίωσή τους ε, και για την εξέβρεση εργασίας, αλλά και για τη σταθεροποίηση, της, σταθεροποίησή τους στην αγορά εργασίας, νομίζω ότι είναι ε, ε, πάρα πολύ έντονο ως εμπόδιο για να μπορούμε να πούμε ότι θα αυξηθεί η συμμετοχή των νέων γυναικών. Αν σε αυτό το άγχος και το φόβο προσθέσουμε και τη φροντίδα στην ευθύνη του νοικοκυριού, δηλαδή παιδιά και εξαρτημένα μέλη, νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλες τις δυσκολίες συμμετοχής των νέων γυναικών στην πολιτική ζωή. Άρα νομίζω είναι αναγκαίο να λάβουμε μέτρα και πολιτικές ε, που θα αφορούν τη ρύθμιση στην αγορά εργασίας, την καλυτέρευση των συνθήκων ε, εργασίας, αλλά και τη βελτίωση του χάσματος στους μισθούς μεταξύ ανδρών και γυναικών. Θα πρέπει αυτό να μας απασχολήσει και θα πρέπει επίσης να μας απασχολήσει και η κατανομή της φροντίδας και των εθνών στον οικοκυριό. Και εδώ θα ήθελα πραγματικά να επισημάνω την αναγκαιότητα αύξησης των δομών ε, της φροντίδας των παιδιών και των εξαρτημένων μελών, καθώς και τις πολιτικές κινήτρων για τη χρήση των γονικών αδειών από τους δύο γονείς. Και ίσως, ε, είπα και προηγούμενα στην, ομιλία μου, ε, στην προηγούμενη ομιλία, ότι πρέπει να δούμε ε, στοχευμένες πολιτικές και για τις χώρες του Νότου όπου για ένα πολύ μεγάλο διάστημα η οικογένεια να πλήρωνε το κράτος πρόνοιας, νομίζω ότι πρέπει να δούμε κάποιες στοχευμένες, παρότι σήμερα έχει εξελιχθεί, δεν υπάρχει αυτό σε μεγάλο βαθμό, να δούμε πώς θα στοχεύσουμε πολιτικές ενίσχυσης των συγκεκριμένων δομών των κοινωνικών υπηρεσιών. Ε, άφησα τελευταίο χωρί να είναι ε, καθόλου, είναι πάρα πολύ σπουδαίο την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων σε όλα τα πεδία πολιτική. Ε, και νομίζω ότι η πρόοδο στην ισότητα των φύλων ε, πρέπει να, ε, τις, οι νέες κοπέλες να μπορούμε με στο, θεσμικά και στοχευμένα μέτρα να έχουμε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των νέων γυναικών για να, και εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουν ε, τα έμφυλα στερεότυπα και τις προδιαγραμμένους, προδιαγραμμένους έμφυλους ρόλους. Πρέπει δηλαδή σε όλες τις πολιτικές και τις οργανωσιακές πρακτικές να ενσωματωθεί η σκοπιά του φύλου και η επικέντρωση στην άρση των έμφυλων στερεοτύπων. Βασικές πολιτικές σε συνδυασμό με ενίσχυση της δημόσιας διαβούλευσης και των πολιτικών πρωτοβουλειών σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής και εδώ αναφέρουμε ιδιαίτερα στα ΜΜΕ. Αυτά, αυτά πρέπει να, είναι, ε, να, να μπορούν να μεταφραστούν σε πολιτικές από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν θέλουμε να πούμε ότι θα μπορούμε να συμβάλλουμε στο να μπορούν να συμμετέχουν περισσότερο οι νέες γυναίκες στην πολιτική. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Θελερίτη. Η κυρία Κλίφορντ από την Ιρλανδία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι εδώ και σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Άκουσα με ενδιαφέρον την ε, συζήτηση για την απόσταση των αμοιβών μεταξύ των φύλων, που είναι και ένα σημαντικό εμπόδιο για τη συμμετοχή των γυναικών. Και το να έχουν στη διάθεσή τους χρηματικούς πόρους οι γυναίκες είναι πολύ σημαντικό. Οι ποσοστώσεις έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο στην Ιρλανδία στις τελευταίες γενικές εκλογές, δηλαδή το 2016, που ήταν η πρώτη φορά, η πρώτη ευκαιρία δηλαδή που εφαρμόσαμε τη σχετική νομοθεσία με πολύ καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή μπήκαν περισσότερες γυναίκες στο κοινοβούλιο μας. Καμιά φορά όμως η πρόοδος αυτή ανακόπτεται. Χρειάζεται προσοχή. Τα πολιτικά κόμματα οφείλουν όχι μόνο να επιλέγουν γυναικείες υποψηφιότητες στις εκλογές, αλλά και να τους δώσουν και την απαραίτητη χρηματική υποστήριξη, ώστε να μπορέσουν να διεξαγάγουν αποτελεσματικές εκστρατείες είναι επίσης λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό. Και το δίκτυο των mentor είναι πολύ σημαντικό για τις νέες γυναίκες υποψήφιες. Δεν έχει δηλαδή η γυναίκα κάποιον με τον οποίο να μπορεί να έχει μια σχέση παροχής συμβουλών. Μία τριετία πριν να εκλεγώ βουλευτή ήταν πολύ σημαντικό που είχα τι συμβουλέ από τη γυναίκα που προηγήθηκε. Και είναι σημαντικό και για τι γυναίκε που έρχονται μετά από μα παρόλο που είναι απαιτητικό ό,τι αφορά τον χρόνο μα, είναι σημαντικό να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τι νεότερες αδελφέ μα στα κόμματα. Θέλω να μιλήσω λίγο, αν με επιτρέπετε, για το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν οι γυναίκες στην πολιτική. Άκουσα με ενδιαφέρον την εκστρατεία του ότι η ευρωβουλευτή μου είναι όπω εγώ. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για μα, ω γυναίκε πολιτικού να μπορέσουμε να πούμε στον κόσμο ότι δεν είμαστε τίποτε εξαιρετικές περιπτώσεις, ούτε είμαστε τέλειες, διότι καμιά φορά οι γυναίκες που εμπλέκονται στην πολιτική τις κάνουν ανδριάντες και αυτό είναι, βάζει πολύ ψηλά τον πύχη σε άλλε γυναίκε για να μπουν στην πολιτική, διότι αυτέ έχουν την αίσθηση, κοιτάξτε εγώ δεν είμαι τόσο καλή, δεν έχω όλα αυτά προσόντα, Πώ θα μπω στην πολιτική. Πρέπει λοιπόν να, δούμε, να πούμε και εμεί ότι έχουμε και εμεί προκλήσει στην πολιτική μα ζωή και εμεί δεν τα ξέραμε όλα όταν αρχίσαμε, αλλά μαθαίνουμε διαρκώ πάνω στη δουλειά όπω λένε. Καμιά φορά αισθάνομαι ότι το φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον και η συμβολή του καμιά φορά υπερτιμώνται. Εγώ ήμουν δικηγόρος πριν να μπω στην πολιτική. Και εκεί το περιβάλλον δεν είναι φιλικό για τις γυναίκες, ούτε για τις οικογένειες. Και η μετακίνηση των ευθυνών για την οικογένεια πρέπει να παίξει και αυτή ένα ρόλο. Όταν κατέβηκα για πρώτη φορά σε εκλογές, ήμουν έγκυος στο πρώτο μου παιδί και την έχασα, Τι έχασα ότι τις εκλογές. Πολλοί άνθρωποι με καλή θέληση μου είπαν καλύτερα που δεν εκλέχθηκες γιατί δεν θα προλάβαινες και το παιδί και την πολιτική. Εγώ όμως δεν την άκουσα τη συμβουλή αυτή, επέμεινα, κατέβηκα στις επόμενες εκλογές και ευτυχώ εκλέχθηκα. Νομίζω ότι πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το συνεχές αφήγημα ότι η πολιτική δεν είναι κατάλληλη για τις γυναίκες. Υπάρχουν κάποια στοιχεία εκεί, αλλά καμιά φορά, ξαναλέω, υπερτιμώνται και τελικώ αποβαίνουν τροχοπέδε και εμπόδια για την συμμετοχή των γυναικών. Thank Ευχαριστώ. Η κυρία Ταμπάρη από την Πορτογαλία κάνει την τελευταία παρέμβαση. Σα ευχαριστώ. Θα μιλήσω στα πορτογαλικά. Ε, πράγματι, η συμμετοχή στην πολιτική ζωή των νεαρών ε, γυναικών είναι δύσκολο και ακόμα πιο δύσκολο είναι ο συνδυασμό τη ιδιότητα τη γυναίκα με την ιδιότητα τη μητέρα. Δεν είναι λοιπόν ε, πάντοτε δυνατό να υπάρξει αυτή η συμμετοχή. Αντιμετωπίζουν δυσκολίε και εγώ όταν ήθελα και ήμουν υποψήφια για, ως βουλευτής στο Εθνικό μας Κοινοβούλιο ήμουνα τρεις μήνες έγκυο και συχνά άκουγα από ε, πολλούς ε, ε, συναδέλφους και πολλούς ανθρώπους που έλεγαν ότι αχ τώρα θα χρειαστεί να μετακομίσεις δηλαδή προς τη Λισαβόνα επειδή έχεις κλαιγή και πώς θα το κάνεις με παιδί και ούτω καθεξής. Δηλαδή πραγματικά αυτή η αντιμετώπιση μας δημιουργεί δυσκολίες στην πολιτική μας ζωή. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε πως είναι δυνατό να βελτιώσουμε τον κόσμο και είναι δυνατό να αλλάξουν τα πράγματα και όπως ήδη υπόθηκε από προηγούμενη ομιλήτρια, όταν ε, μια γυναίκα ε, ε, εισέρχεται στον πολιτικό κόσμο, αλλάζει η ίδια. Αλλά όταν έχουμε πολλέ γυναίκε οι οποίε εισέρχονται στον πολιτικό κόσμο, αλλάζει ο πολιτικό κόσμο. Άρα λοιπόν θα βλέπουμε ότι το γεγονό ότι βλέπουμε μια πιο δίκαια ε, εκπροσώπηση τη σήμερα ημέρα οφείλεται ακριβώ και στην υψηλότερη εκπροσώπηση ε, των γυναικών ε, στην πολιτική ζωή. Και ένα ακόμα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι η ιδιότητα τη μητρότητα και τη πατρότητα, στο οποίο αναφέρθηκε η Τζάκη. Δηλαδή, δεν θέλουμε να έχουμε να παραγνωρίζουμε ούτε τη μητρότητα ούτε την πατρότητα. Εκείνα τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να λαμβάνουμε θα πρέπει να αντιμετωπίζουν αυτέ τι ιδιότητε ω ιδιότητα του γονέα γενικότερα, χωρί διάκριση. Και ακριβώ η υποχρέωση που βαρύνει κυρίως τις γυναίκες ε, ε, για να ε, φροντίζουν τα παιδιά είναι ένα εμπόδιο το οποίο έχει υπάρξει και για, τις, για τη συμμετοχή στην πολιτική ζωή των γυναικών και των εργαζομένων γυναικών αλλά και στην αγορά εργασίας. Άρα λοιπόν το μήνυμα που θα ήθελα να περάσω είναι ότι βλέπουμε ε, λαμβάνονται κάποια μέτρα. Για παράδειγμα, είδαμε και την νομοθεσία που εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα στην ε, Ισπανία, δηλαδή την ίδια άδεια μητρότητα και πατρότητα ε, για του γονεί. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε την δυνατότητα ακριβώ ε, να παρέχουμε ε, την ίδια δυνατότητα. Δηλαδή όταν κανεί εξετάζει έναν υποψήφιο για μια θέση εργασίας ε, να εξετάζει όλα τα ζητήματα ανεξαρτήτω του αν πρόκειται για άνδρα ή για γυναίκα. Δηλαδή να μην η άσκηση αν θέλετε όσων σχετίζονται των υποχρεώσεων με την μητρότητα να μην αποτελεί εμπόδιο για την συμμετοχή σε αυτή τη ζωή. Δηλαδή να μην υπάρχει δυσμενή διάκριση, διαχωρισμό τη γυναίκα στο πλαίσιο τη αγορά εργασία Και κάτι τέτοιο βέβαια έχει ε, και ε, θετικό αντίκτυπο στην ίδια τη μητρότητα. Γιατί έχουμε μια Ευρώπη η οποία γυράσει όλο ένα και περισσότερο. Άρα λοιπόν θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο της υπογεννητικότητας ε, ακριβώς και με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να δώσουμε τη δυνατότητα στις νεαρές γυναίκες να έχουν περισσότερα παιδιά. Και όπως αναφέρθηκε ήδη από την συνάδελφο που ενέβη από την ε, ε, Πορτογαλία. Τέτοιου είδου πολιτικέ θα πρέπει να στοχεύουν στο να έχουν τη δυνατότητα γυναίκε να έχουν παιδιά και μάλιστα όσα παιδιά επιθυμούν. Θα πρέπει να δώσουμε τα κατάλληλα κίνητρα, τι ε, καλύτερε συνθήκε εργασία και δυνατότητε εργασία για τι νεαρέ γυναίκε και θα πρέπει να έχουμε καλύτερη κατανομή των διαφορετικών υποχρεώσεων και σε οικογενειακό επίπεδο μεταξύ ανδρών και γυναικών. θα πρέπει δηλαδή να κάνουμε και το σχετικό διάλογο σε ό,τι αφορά την άδεια μητρότητα, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τι γυναίκε, αλλά να κάνουμε γενικότερο διάλογο σε ό,τι αφορά άδεια γονική ε, μητρότητα και πατρότητα, ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε ε, συνέχεια στα όσα είχα αναφερθεί σε μια προηγουμένη έκθεση και αναφέρθηκε εδώ από μια πρώην Ευρωβουλευτή, όπου αναφέρεται ακριβώς η ανάγκη λήψη μέτρων και χορήγηση άδεια και μητρότητα αλλά και πατρότητα σε όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το μήνυμα που ήθελα να περάσω από την πλευρά μου σήμερα το πρωί. Σα ευχαριστώ πολύ. Σας Ευχαριστώ κυρία Ταβάρες. Πριν δώσω το λόγο στις ε, συντρόφους μας για να απαντήσουν, θα ήθελα να πω το εξή, ότι όταν μιλάμε για την πολιτική συμφιλίωση, αυτή δεν είναι πολιτική γυναικών. Εμείς μια ζωή την περνάμε συμφιλιώνοντας. Ε, θυμάστε τις α, ε, γιαγιάδες μας, τις μητέρες μας που δούλευαν μέσα και έξω από το σπίτι. Ε, πρέπει να δούμε ότι και στο χώρο εργασία οι άντρε είναι η συντροφή μας. Ε, γι' αυτό λοιπόν στο Κοινοβούλιο είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε τη συμφωνία που φτάσαμε με το Συμβούλιο για τη γονική άδεια. ούτω ώστε να χωρίζεται η γονική άδεια στους πατέρες και στις μητέρες. Ε, παλιά, στην αρχή μάλλον ξεκινήσαμε τις, τους τέσσερις μήνες αυτής της γονικής άδειας, ε, όπου η θέση ήταν ότι θα ήταν μη μεταφερόμενε από τον πατέρα στη μητέρα. Τώρα λέμε ότι δύο μήνε δεν μεταφέρονται, είναι για τον ένα και οι άλλοι δύο μπορούν να περάσουν από τον ένα στον άλλον γονιό. Ε, είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί αυτή η συνδιαλλαγή, γιατί θα μας εξασφαλίσει την ισότητα των ευκαιριών και την ίση πρόσβαση ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας. Για να μην ξαναακούσουμε την ερώτηση από εργοδότη προς γυναίκα που έχει την κατάλληλη ηλικία για να γίνει μητέρα, θέλεις να γίνεις μητέρα ή όχι. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην Ινέση για να απαντήσει. Ινέση Σουμπέρ. Ε, ευχαριστώ. Ε, σύντομα θα απαντήσω γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μα. Ε, θα ήθελα και εγώ να επαναλάβω αυτή την έκκληση ότι όταν δηλαδή αναφερόμαστε στην συμμετοχή στην πολιτική ζωή και γενικότερα στην, στα κοινά θα πρέπει να εξετάζουμε ή να δίνουμε έμφαση στις γυναίκες εκείνες οι οποίες έχουν ήδη τις δυνατότητες να συμμετάσχουν στην πολιτική ζωή αλλά σε όλες τις γυναίκες. Δηλαδή όταν αναφερόμαστε στην υψηλότερη συμμετοχή ε, των γυναικών, για παράδειγμα στα Εθνικά Κοινοβούλια εδώ, θα πρέπει πάντοτε να εξετάζουμε την ε, ανισότητα που υφίστανται οι γυναίκε γενικότερα σε ό,τι αφορά την ε, πρόσβαση σε αυτή την πολιτική ζωή και στην κοινωνία των πολιτών. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα, για να τελειώσουμε αυτό το κομμάτι, θα δώσω το λόγο στην Καρίμα που θα κάνει και τις τελικές παρατηρήσεις. Καρίμα. Yes, it's very unusual to have two Karimas in the panel. Με δύο Καρίμα. Δύο γυναίκες που λέγονται Καρίμα είναι πολύ ασυνήθιστο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση. Συμφωνώ με τη συνάδελφο από την Ελλάδα για το θέμα της πρόοδου. Ελπίζω να προχωρήσαμε κάπως, γιατί μετά από πέντε χρόνια αισθάνομαι ότι έχουμε κάνει κάποια πράγματα, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να κινηθούμε με, περισσότερο, με πιο γοργό βήμα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο και θα πρέπει σε μικρό χρονικό διάστημα να κάνουμε πολλά, να πετύχουμε την ισότητα των φύλων, να συμμετέχουν ε, στις ε, αποφάσεις οι γυναίκες ε, σε όλα τα επίπεδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σαΐ. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στην πρόεδρο της Επιτροπής ε, Μεταφορών από τους Πράσινους, την ε, Ευρωβουλευτή κυρία Καρίμα Ντελή. Θα μιλήσω γαλλικά. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ τη συνάδελφο. Είναι φανταστική γιατί η Επιτροπή αυτή γυναικών και δικαιωμάτων των γυναικών γίνεται όλο και πιο παρούσα, όλο και πιο ορατή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε ευχαριστώ λοιπόν, ε, γιατί πρέπει και εμείς να βάλουμε το λιθαράκι μας εκεί που πρέπει. Εγώ είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και ποτέ δεν υπήρχε πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών επί 40 χρόνια πριν από μένα. Είναι σκανδαλώδες. Όταν έφτασα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήμουν πάρα πολύ μικρή, πολύ νεαρή. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και ο πολιτικό κόσμος είχε διαμορφωθεί από τους άντρες για τους άντρες. Έφτασα λοιπόν νεαρότατη, θα σας πω τώρα και μια μικρή ιστορία και μετά θα φτάσω στο συμπέρασμά μου τότε ο κύριος Μπούζεκ ήταν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ ήμουν στην ε, γαλλική αντιπροσωπεία και είπε σε ένα δείπνο, καλημέρα σε όλους τους ε, ευρωβουλευτές, φτάνει μπροστά μου και λέει «Τι ωραίο είναι αυτό το επάγγελμα που κάνετε». Τον κοιτάω λοιπόν και μου λέει «Πόσες γλώσσες μιλάτε». Του λέω «Τρεις». «Αχ, θα ήθελα και εγώ να είμαι διερμηνέας», είπε ο κύριος Μπούζεκ. Και του λέω, το απαντάω, δεν είμαι διερμηνέας, είμαι και εγώ βουλευτής. Αυτό είναι το πρόβλημά μας ακριβώς. Γιατί στο ασυνείδητό του είμαστε νεαροί, δυναμικοί, γυναίκα, αλλά δεν είμαστε στην πολιτική. Ε, όχι κυρία μου, μπορούμε να είμαστε και πολιτικές, πολιτικοί. Αυτή είναι η φραγμή, αυτά είναι τα εμπόδια. Όλοι μας λένε είναι δύσκολο μια γυναίκα να είναι πολιτικός, να δουλεύει 12 ώρες τη μέρα, γιατί πρέπει να είμαστε πάνω απ' όλα καλή μητέρα, καλή εργαζόμενη, επικεφαλής επιχείρησης, πρέπει να είμαστε καταπληκτικές νοικοκυρές, ε. αλίμονο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε. Και επίσης πρέπει να είμαστε και καλή σύζυγος. Και η κοινωνία μάλιστα μας ενοχοποιεί, μας κάνει να αισθανόμαστε ένοχοι. Γιατί οι νεαρές γυναίκες δεν θέλουν να κατέβουν στην πολιτική. Γιατί, και το είπατε εσείς κυρία μου, γιατί υπάρχει μια σύγκρουση σε κοινωνικό επίπεδο. Να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Εγώ είμαι από μια εργατική οικογένεια. 13 παιδιά είχαν οι γονείς μου, είμαι η ένατη στη σειρά. Στις ε, τάξεις αυτές, τις εργατικές τάξεις, Κανένα δεν θεωρεί ότι πρέπει να κάνει ένα κορίτσι να κατέβει στην πολιτική, αλλά αντίθετα πρέπει να βρει δουλειά. Αυτά είναι στο μυαλό όλων από τα εργατικά στρώματα. Αυτά τα εμπόδια πρέπει να τα σπάσουμε. Αυτούς τους φραγμούς, αυτήν την οτροπία. Επομένως, πρέπει να υπάρχει μισθολογική ισότητα, γιατί είναι σκανδαλώδες το αντίθετο. Ε, στην Επιτροπή απασχόληση, Αγαπητοί συνάδελφοι, όσοι είστε εκεί, ε, πόσα ψηφίσματα δεν έχουμε υιοθετήσει, ε, πόσε φορέ δεν έχουμε πει να τελειώσει πια η διακριτική μεταχείριση. Θέλουμε ίσα δικαιώματα ανάμεσα στου άνδρες και γυναίκε. Αυτό είναι το τμήμα των αξιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πράξη όμω, πού είμαστε, πού έχουμε φτάσει, όταν κοιτάζω την τελευταία έκθεση του Οικονομικού Παγκόσμιου Φόρουμ ε, μία μελέτη για 149 χώρες δείχνει ότι με αυτό το μισθό, μισθολογική, με αυτό το ρυθμό, η μισθολογική ισότητα, αν συνεχίσουμε ακριβώς έτσι, θα πετύχουμε αυτή την ισότητα σε 108 χρόνια. Σε 108 χρόνια θα, θα πετύχουμε την μισθολογική ισότητα. Ε, δεν θέλω να περιμένουμε 108 χρόνια για να πετύχουμε αυτή την ισότητα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να περάσουμε όχι μόνο τους νόμους, γιατί μοιάζουν όμορφοι, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζονται. Όταν δεν εφαρμόζονται, τι χρειάζεται, κυρώσει. Θα πρέπει να τιμωρούμε με κυρώσει την μισθολογική ανισότητα. Αν κάνουμε τα ίδια πράγματα με τον άντρα, θα πρέπει να παίρνουμε τα ίδια λεφτά. Τελεία. Επίσης, η εκπροσώπηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είδαμε πολλέ φορέ να μιλάμε για την εκπροσώπηση στα διοικητικά συμβούλια για την εκπροσώπηση των γυναικών στον επιχειρηματικό κόσμο, στις υψηλές θέσεις. Έχουμε σχετικούς νόμους, σχετικούς κανόνες. Εφαρμόζονται όλα αυτά. Όχι. Όταν διαβάζουμε λοιπόν για, την, για τον πολιτικό στίβο, ας πούμε, να υπάρχουν νόμοι για την ισότητα, για να μας ανοίξουν οι πόρτες. Αυτοί οι νόμοι βοηθάνε. Ανοίγουν οι πόρτες και είμαστε περισσότερες γυναίκες τώρα. Ε, η παρουσία των γυναικών όμως δεν θα πρέπει να υπάρχει μόνο στην πολιτική, θα πρέπει να υπάρχει και στο συνδικαλισμό, στις οργανώσεις, στι επιχειρήσεις, παντού. Εδώ δώσαμε μάχη για να πετύχουμε την άδεια. Τη γονική άδεια δηλαδή. Ε, και οι άντρες ακόμη μερικές φορές είπαν ότι θέλουν και αυτοί δικαίωμα σε αυτή την άδεια και σπρώξαμε ούτω ώστε να πετύχουμε αυτό το μοίρασμα. Γιατί υπάρχουν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων που ήταν αντίθετοι, γιατί λέγανε ότι θα κοστίσει πάρα πολύ αυτό. Είναι αδιανόητο και παλαβό το 2019 να λέμε τέτοια πράγματα, ότι θα μας κοστίσει πολύ. Το γεγονός ότι αύριο, μεθαύριο, οι άντρες ε, θα πάρουν άδεια γονή για τα παιδιά τους, αυτό θα είναι βολικό και, και επικερδές για το ζευγάρι, γιατί η γυναίκα θα μπορέσει να βρει δουλειά. Για να μην είμαστε παθητικά όργανα στην κοινωνία, εμείς οι γυναίκες. Πρέπει να προχωρήσουμε και εκεί. Λοιπόν, τελευταίο πράγμα που θέλω να σας πω. Νομίζω ότι οι γυναίκες είναι λιγάκι υποταγμένες και αντιμετωπίζουν φραγμούς που δεν τους ονοματίζουμε. Δηλαδή, τα δεχόμαστε όλα αυτά που μας επιβάλλουν, το είπαν κάποιοι συνάδελφοι. Δεχόμαστε αυτού του ψυχολογικού φραγμού, αυτού του κοινωνικού φραγμού. Ε, λέμε ίδιοι στον εαυτό μα. Α, δεν έχω αρκετό χρόνο για να κατέβω στην πολιτική, γιατί είναι δύσκολο αυτό. Δεν μπορώ να οργανώσω το χρόνο μου για να το κάνω. Και κυρίω. Θα μου δυσκολεύσει πάρα πολύ τη ζωή. Μας βάζουν φραγμούς και μας λένε ότι δεν έχουμε την ικανότητα να επιβληθούμε, να παίξουμε ηγετικό ρόλο, ότι δεν έχουμε σωστή κρίση, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην κρίση μας και τον εαυτό μας. Οι άρενες συνάδελφοι που είναι εκεί τμήμα του κατεστημένου είναι πολύ καλύτεροι για τις θέσεις. Τα είπατε όλα αυτά, έτσι. Υπάρχουν φραγμοί που επιβάλλει η κοινωνία στις γυναίκες. Και μερικές φορές οι γυναίκες το καταπίνουν αμάσιτα, δεν καταλαβαίνουν καν ότι το έχουν αποδεχτεί. Γι' αυτό λοιπόν εγώ λέω ότι έχουμε φτάσει στο 2019. Λίγες, μέρες, λίγες ώρες μας χωρίζουν από την ε, Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Ακούστε εσείς οι άντρες, πρέπει να μας έχετε εμπιστοσύνη. Πρέπει να τολμήσουμε εμείς οι γυναίκες, να μπούμε στην πολιτική, να έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, να δείξουμε ότι έχουμε τα ίδια προσόντα με τους άντρες, να πούμε ναι σε ένα κόσμο που θα λαμβάνει υπόψη όλες τις γυναίκες. Ας τολμήσουμε να πούμε όχι στους ρόλους που θέλουν να μας κολλήσουν. Και εσείς κύριοι μου, για να μην σας ξεχάσουμε, πιέστε τις γυναίκες σας, τους φίλους σας, τα κορίτσια σας, τις μανάδες σας, να έρθουν στο πλευρό μας, να κινητοποιηθούν. Γιατί και εσείς πρέπει να μας βοηθήσετε. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι δεν τα καταφέρνουμε μόνες, από μόνες, πρέπει και εσείς να μιλήσετε, να εκφραστείτε δημόσια για το ποιο είναι το όραμά σας για μια μελλοντική κοινωνία ισότιμη, την οποία θα χτίσουμε μαζί. Ευχαριστώ. Muchas, muchas gracias. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Ντελή. Τελειώσαμε με μεγάλο πάθος, με μεγάλο ζήλο αυτό το πάνελ. Με μεγάλη χαρά το μοιράστηκα μαζί σας. Και τώρα ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ε, Δικαιωμάτων των Γυναικών, ο κύριος ε, Πιμέντα και μετά η κυρία Μογκερίνη, για να τελειώσουμε εδώ αυτή την εκδήλωση. Muito bem. Eh, πολύ ωραία. Ε, συνεχίζουμε λοιπόν τις εργασίες μας και ε, αναμένουμε δεν είπατε εκπρόσωπο τη Φεντερίκα Μοντερίνη ακόμα για να ακούσουμε και μια τελική παρέμβαση από τη δική της ε, πλευρά. Ελπίζουμε λοιπόν να καταφέρει να καταφτάσει. Μετά λοιπόν, μετά από αυτή την, ε, τον, τον, την παρέμβαση γεμάτη πάθος από την πλευρά της συναδέλφου Κάρη Μαντέλη, είναι δύσκολο για μένα να προσθέσω νέα στοιχεία ε, σε αυτή τη συζήτηση μετά και από όλες τις υπόλοιπες παρεμβάσεις και τα όσα ακούσαμε ε, στη σημερινή συζήτηση. Δηλαδή είναι δύσκολο πραγματικά να προσθέσω κάτι καινούριο. Άρα λοιπόν, εκείνο που θα προσπαθήσω να κάνω είναι να αντλήσω κάποια συμπεράσματα από τα όσα υπόθηκαν σήμερα εδώ και να σημειώσω κάποια στοιχεία. Η Επιτροπή λοιπόν αυτή εδώ έχει αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό φόρουμ για να κάνουμε κάποιες σκέψεις σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ισότητας των φύλων και το ε, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε λύσεις για το μέλλον. Όμως ε, όπως ακούσαμε και στο πλαίσιο των διαφόρων παρεμβάσεων, είναι δύσκολο να το εξετάσει κανείς αυτό χωρίς ε, την ε, οπτική γωνία εκείνη η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε ένα πολύ διατομιακό αν θέλετε στοιχείο. Και αυτό είναι το γεγονός ότι η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή έχει να κάνει με, ένα, με μια σειρά από περαιτέρω στοιχεία. Δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με την πολιτική ζωή, έχει να κάνει με την οικονομική ζωή και όλες εκείνες τις διαφορές και τις δυσμενείς διακρίσεις που υφίστανται συστηματικά οι γυναίκε. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε, να οικοδομήσουμε μια προοδευτική και δίκαιη ε, κοινωνία, εάν δεν λάβουμε υπόψη μας όλες αυτές τις διαφορετικές διαστάσεις ε, τη ζωή. Και όπως αναφέρθηκε εδώ, υπάρχει ακριβώς μια τέτοια ε, σύνθεση εδώ που αναδεικνύεται με βάση όλα αυτά τα στατιστικά στοιχεία και τα δεδομένα που έχουμε ε, που καταδεικνύουν ε, την ε, ένδυα της δυσμενή διακρίση στην αγορά εργασία, τη διακρίση και τα εμπόδια που δημιουργούνται λόγω τη μητρότητα και ούτω καθεξή. Άρα λοιπόν, οι στρατηγικέ οι οποίε υιοθετούνται, η νομοθεσία που θεσπίζεται, αποτελούν όλε τι προσπάθειε και απόπειρε να αντιμετωπιστούν αυτέ οι ανισότητες και διακρίσει όμω, όπω κατέστησε σαφές ουσιαστικά σε όλε τι παρεμβάσει που ακούσαμε, Παρότι όλα αυτά λοιπόν προβλέπονται, θεσπίζονται νομοθετικά, οι βασικές δηλαδή αρχές, οι οποίες αποτελούν ε, πυλώνες αν θέλετε για την ε, καλή λειτουργία ενός δημοκρατικού πολίματος, δεν βλέπουμε την εφαρμογή του στην πράξη, στην, στην καθημερινή ζωή. Είδαμε πρόσφατα ένα ψήφισμα από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ακριβώς σε σχέση με αυτό το ζήτημα, δηλαδή της επαναχώρησης των δικαιωμάτων των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μία σειρά από στην αγορά εργασίας, ε, στο θέμα της μητρότητας, στα θέματα παιδείας. Ε, σε ό,τι αφορά την ε, βία εις βάρος των γυναικών, που αποτελεί και ένα ζήτημα επίκαιρο τη σημερινή ημέρα για τους πλέον θλιβερούς λόγους. Και έτσι λοιπόν αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν νόμοι που μάλιστα έχουν και μεγάλη εμβέλεια, αλλά δεν εφαρμόζονται στην πράξη. Άρα λοιπόν διατρέχουμε τον κίνδυνο να ε, υπάρξουν εδώ πολλές δηλώσεις πρόθεσης, να υπάρξουν πολλά νομοσχέδια, αλλά να μην υπάρξει συγκεκριμένη ανάληψη δράσης, είτε σε επίπεδο εθνικών κυβερνήσεων, είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή δεν υπάρχει ο κίνδυνος του να μην υπάρξει πραγματική εφαρμογή στην πράξη και πραγματικές αλλαγές Αλλαγέ δηλαδή στην καθημερινή ζωή. Και είδαμε και ένα διάγραμμα εδώ σε μια παρουσίαση η οποία, το οποίο κατέδειχνε την, εξελίξει τις εξελίξεις από το 2005 έως το 2015. Είδαμε λοιπόν ότι στην ε, ε, πλειοψηφία των κρατών μελών υπήρξαν ε, κάποιες βελτιώσεις, αλλά πραγματικά οριακές, οριακές βελτιώσεις. Και εδώ βέβαια τίθεται και το ζήτημα της ε, συμφιλίωσης μεταξύ της οικογενειακής και της επαγγελματική ζωής και το, και το ζήτημα των σχολιών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε ό,τι αφορά την, ακριβώς την απουσία της ε, προστασίας της εργασίας, της προστασίας της μητρότητας ε, ε, και μία σειρά από διακρίσεις και ανισότητες που ουσιαστικά οδηγούν την γυναίκα στο να αποκλειστεί από την αγορά εργασίας. Και αυτό βέβαια με τη σειρά του οδηγεί στην διαιώνιση της ανισότητας αυτού του φαύλου κύκλου, γιατί υπάρχουν ε, και μελέτες οι οποίες καταδεικνύουν ότι σε 200 χρόνια από τώρα θα έχουμε καταφέρει να φτάσουμε σε μια πραγματική ισότητα και δεν μπορεί, δεν μπορεί κάτι τέτοιο να αποτελεί το δικό μας ε, στόχο, τη δική μας άγουσα. Άρα λοιπόν, εκείνο που δεν συμβαίνει στην πράξη είναι να εφαρμόζεται εκείνο που προβλέπεται στην ομοθεσία και στην πραγματικότητα. Και εδώ βέβαια αναφέρομαι και σε ένα ζήτημα το οποίο είναι θεμελιώδη σημασία και αναφέρθηκε από πολλού, δηλαδή ε, τη μισθολογική ισότητα. Και η, αναφέρθηκε ήδη από κάποιον ότι ουσιαστικά υπήρξαν 11 διαφορετικοί νόμοι οι οποίοι ε, θεσπίστηκαν ακριβώ για να διασφαλιστεί η μισθολογική ισότητα, χωρί τελικά να ισχύει στην πράξη. Γιατί τελικά ε, οι νόμοι αυτοί δεν μεταφράζονται στην ε, συγκεκριμένη ανάληψη μέτρων για την εξασφάλιση ακριβώ ε, της εξάλληψης ε, του μισθολογικού χάσματος. Ε, επίσης κάτι άλλο ε, που θα ήθελα να αναφέρω εδώ ε, είναι ότι δεν θα πρέπει να αποτελεί αυτό σκοπό η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή. Θα πρέπει δηλαδή να δημιουργήσουμε όλες τις απαραίτητες συνθήκες για την συμμετοχή στην πολιτική των ε, γυναικών επί ίσης όρης, αλλά μία τέτοια διαδικασία θα πρέπει να συνοδευτεί από μία αντίστοιχη αλλαγή όλων εκείνων των συνθήκων, όλων των παραμέτρων οι οποίες εμποδίζουν ε, την ε, συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική και οικονομική ζωή. Δηλαδή, αναφέρομαι εδώ σε αλλαγές οι οποίες θίγουν ακόμα και την προσωπική ζωή της γυναίκας. Και εδώ αναφέρομαι για παράδειγμα στο ζήτημα της επισφαλούς εργασίας, της απορρίθμισης των ωραρίων εργασίας, στο ζήτημα ε, της ολοένα και αυξανόμενης ένδυας γιατί ας μην ξεχνούμε ότι ε, σχεδόν το 1 τέταρτο της, ε, του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, διαβεί σε συνθήκες κινδύνου, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Και βέβαια ένα σημαντικό κομμάτι αυτού του 1 τετάρτου είναι γυναίκες. Είναι γυναίκες. Και η, αυτή λοιπόν η κατάσταση της φτώχειας και η κατάσταση της επισφαλούς εργασίας κυρίως αφορά γυναίκες ή για παράδειγμα το ζήτημα της ε, φροντίδας ε, συγγενών. Είναι κάτι το οποίο οδηγεί τελικά πολλές ε, γυναίκες από το να απομακρυνθούν από την αγορά εργασίας ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν διαφορετικές εναλλακτικέ δεν δίνονται δυνατότητες αυτές τις γυναίκες από την ίδια την κοινωνία. Επειδή επίσης αναφέρθηκε το ζήτημα της προστασίας της μητρότητας και το γεγονός ότι σε πολλά κράτη-μέλη δεν είναι εγγυημένη η προστασία αυτής της μητρότητας. Και αναφερθήκαμε στο πώς αυτό δημιουργεί προβλήματα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, πολλέ φορέ βλέπουμε να έχει κατοχυρωθεί νομοθετικά η προστασία τη μητρότητα, αλλά συχνά πολλέ κυβερνήσει ή μάλλον συγγνώμη, πολλέ γυναίκε ε, παρετούνται, αν θέλετε, από την άσκηση αυτού του δικαιώματο του ακριβώ επειδή βρίσκονται ε, αντιμέτωπες με απειλές του να απολέσουν τη θέση εργασίας τους. Εάν δηλαδή αξιώσουν την, ε, το να μπορέσουν να, να, να χάνουν το δικαιώματο τους. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε εδώ όχι περισσότερους νόμους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά συγκεκριμένα μέτρα. Μέτρα τα οποία θα θεσπίσουν στην πράξη, θα εφαρμόσουν στην πράξη τα όσα αξιώσαμε σήμερα το πρωί. Δεν θα επεκταθώ πολύ παραπάνω. Νομίζω πως οι παρεμβάσεις που έγιναν σήμερα εδώ ήταν ε, πολύ συνεκτικές, ε, πολύ συνεπείς ε, και πολύ προσφυείς σε ό,τι αφορά το, την άγουσα που θα πρέπει να ακολουθήσουμε από εδώ και στο εξή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ισότητα των φίλων στο μέλλον και θα κλείσω λέγοντας ότι δεν μπορεί ο αγώνας για την ισότητα μεταξύ των δύο φίλων να περιορίζεται στην, στο να χαιρόμαστε σήμερα την ε, Παγκόσμια Μέρα στις Γυναίκες. Είναι ένας αγώνας στον οποίο θα πρέπει να δίνουμε καθημερινά. Και αυτή την δέσμευση την αναλαμβάνω εγώ προσωπικά για μένα. Και βέβαια αναμένω από όλα τα μέλη της Επιτροπής ε, ΦΕΜΑ αλλά και από την πλευρά όλων των συμμετοχόντων να συμβάλλουν ε, σε αυτή την προσπάθεια. Σε κάτι το οποίο βέβαια είναι όλο και πιο δύσκολο γιατί ενδεχομένως να βρισκόμαστε σε ένα, σε δύο, σε πέντε, σε δέκα χρόνια εδώ και πάλι αξιώνοντας τα ίδια πράγματα τα οποία ε, συζητήσαμε και θέσαμε σήμερα εδώ. Εάν δηλαδή θέλουμε να μετατρέψουμε, να φώσουμε την κοινωνία μας σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, τότε θα πρέπει να περάσουμε στην ε, ανάπτυξη συγκεκριμένων μέτρων. Αυτά από την πλευρά μου τώρα δεν ξέρω αν έχουμε κάποια νέα σε ό,τι αφορά το κατά πόσο θα μπορεί η Επίτροπος να παρευρεθεί εδώ ή όχι. Με ενημερώνουν ότι μέσα σε ένα λεπτό θα βρίσκεται εδώ. Οπότε δείξτε λίγη υπομονή σας παρακαλώ για να ακούσουμε και την παρέμβασή της. Ο πλευρά της κυρίας Μογκερίνη. Από την δική μου πλευρά βέβαια αποχαιρετώ όλους όσους ε, συμμετείχαν από την πλευρά των Εθνικών Κοινοβουλίων και τους ευχαριστώ. και ευχαριστώ όλους όσους ε, παρακολούθησαν τις σημερινές μας εργασίες. Κάνουμε λοιπόν μια πάρα πολύ σύντομη διακοπή αναμένοντας ε, την ε, Επιτροπό Eu pedia só aos presentes que... Θα ήθελα os, os seus lugares. I would call the, the, the, all the, the present to, to return to, to, to their seats. Θα ήθελα όσοι παρευρίσκεστε ακόμα στην αίθουσα να καθίσετε, γιατί καταφτάνει η Επίτροπο, αλλά ενδεχομένω να μην έχουμε διερμηνία. Γιατί οι διερμηνείς ολοκληρώνουν τώρα εδώ το ωράριό του.